Uh, Καλώς ήρθατε στην σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Απασχόλησης. Σας ευχαριστώ για το πολύ ενδιαφέρον και επικοδομητικό απόγευμα που είχαμε χθες. Θα ξεκινήσουμε από το σημείο 6 της ημερήσιας διάταξης. Προϋπολογισμός, εντολή για τον τριμερή διάλογο. Θα έχουμε ανταλλαγή απόψεων με τον εισηγητή της Επιτουσίας Αρμόδιας Επιτροπής, τον κύριο Φερνάντες. Η συζήτηση ακολουθεί συζητήσεις που ήδη έγιναν πάνω στο σχέδιο γνωμοδότησης για την εντολή για τον τριμερή διάλογο για τον προπολογισμό του 2016. Ελπίζουμε ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα προσέλθουν στο μεταξύ δίνω το λόγο στον Γενικό Εισηγητή κύριο Φερνάντες. Παρακαλώ έχετε το λόγο. Euh, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Έρχομαι εδώ για αυτή την ανταλλαγή απόψεων και παρουσίαση, ευχαριστώντας τους συναδέλφους, αλλά και για να καταλάβω τις δικές σας προτεραιότητες, για να έχουμε τον καλύτερο δυνατό προϋπολογισμό. Θυμίζω ότι ήδη στην ορομέλεια της 11ης Μαρτίου είχαμε υιοθετήσει τις κατευθυντήριες γραμμές με τα τρία ε δηλαδή απασχόληση επιχειρήσεις και πάνω απ' όλα μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις όπως και επιχειρηματικό πνεύμα. Δεν ξεχνούμε επίσης την εστερική αλληλεγγύη. Η πολιτική συνοχή είναι σημαντική, αλλά είναι σημαντική, αλλά είναι σημαντική για αυτά τα τρία και ιδιαίτερα την απασχόληση. Την εξωτερική αλληλεγγύη. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τι συμβαίνει γύρω μας. Όπως και τα θέματα ασφάλειας και μετανάστευσης. Τώρα, η βασική μας αρχή είναι ότι το Συμβούλιο και η Κομισιόν θέλει να σεβαστεί τις συμβαστικές λύσεις. Δηλαδή, ότι το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο θα πρέπει να γίνει σεβαστό, ότι οι πληρωμές θα πρέπει να τοποθετούνται στο πλαίσιο της συμφωνίας σύμφωνα με την οποία δεν θα υπερβαίναμε τα 2 δισεκατομμύρια μη καταβληθέντων για το 2016. Και οι πληρωμές είναι συνέπεια των δεσμεύσεων. Είναι λογική συνέπεια των δεσμεύσεων και αυτό θα πρέπει να γίνει σεβαστό. Αλλά σεβόμενοι το πολιτισμό δημοσιονομικό σημαίνει να χρησιμοποιούμε και την ευελιξία. Αποδεχθήκαμε την μείωση λόγω χάρη την ευελιξία. Επομένως και τα περιθώρια μη χρησιμοποιημένων που μπορούν να χρησιμοποιούνται σε επόμενο έτος. Είναι μία από τις καινοτομίες και τα στοιχεία ευελιξίας αυτού του πολυετούς πλαισίου. Όλα αυτά έχουν βεβαίως συνέπειες για τα προγράμματα που μπορούν να βοηθήσουν στην ε, μεγέθυνση για παράδειγμα. Επί του χρονοδιαγράμματος στην Επιτροπή Προεπολογισμού θα υιοθετήσουμε την έκθεση 23 Ιουνίου μετά έχουμε την ορμέλεια του ηλίου μετά έχουμε υποβολή των τροπολογιών μέσα Σεπτεμβρίου υιοθέτηση ενώπιση του ψηφίσματος του Οκτωβρίου μετά ψήφιση των τροπολογιών 28 Οκτωβρίου ψήφιση στην Ολομέλεια 18 Δεκεμβρίου ρωτήσαμε καλά τον ομιλητή συμφιλίωση επομένως στις 27 Μαΐου υπευλήθη για πρώτη φορά και υιοθετήσαμε όπως σας έλεγα σε διοργανική συνάντηση το σχέδιο αυτό των πληρωμών. Και αναφέρομαι στον στόχο να μην έχουμε άνω των δύο δις μη καταβληθέντων σχετικά με τα προγράμματα της περίοδου 7-13. επί των κονδυλίων που μας απασχόλησαν στην Επιτροπή. Είχαμε μια συμφωνία. Αυτά θα έχουν συνέπεια επί του προϋπολογισμού. Προσπαθούμε να μειώσουμε τον αντίκτυπο επί του ορίζοντα 2020 στο ένα δις. Δηλαδή είχαμε περικοπές 6 δις αρχικά, τώρα είναι 5 χρησιμοποίησαμε αυτό το ένα ειδήσιο στα περιθώρια και για το 1α υπάρχει ένα πρόγραμμα καινοτομία ε, και απασχόλησης αυτό θα μπορούσα να πω ότι παραμένει σταθερό σε σχέση με το 15 γιατί δεσμεύσει έχουμε αύξηση 2 εκατομμυρίων και δαπανών 0,5 Μιλώ ε, για, το μηχανισμό μικροχρηματοδότησης κυρίως. Τώρα για το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης Στο σχέδιο προϋπολογισμού έχουμε 165,6 εκατομμύρια δεσμεύσεις και ποσό θα έλεγα εξαιρετικά συντηρητικό 30 εκατομμύρια. Δηλαδή 5 επιπλέον αν συγκρίνουμε με το 15. Για το προσωπικό έχουμε τις μειώσεις. Οι οργανισμοί προτείνουν κατάργηση θέσεων για το Eurofond και για τη ΣΥΝΤΕΦΟ. Τα περιθώρια είναι μειωμένα στο 1α και αυτό έχει αντίκτυπο και για τα προγράμματα πιλότο και τις προπαρασκευαστικές δράσεις, τα οποία δύο περιορίζονται από τον κανονισμό του προϋπολογισμού, όπου έχουμε 100 εκατομμύρια για τις δράσεις και 40 για τα πιλωτικά, 140 σύνολο, αλλά επιπλέον περιορίζονται από τα περιθώρια. Έχουμε πρόβλημα με το 3 όπου δεν έχουμε καθόλου περιθώρια και πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τον μηχανισμό ευελιξίας και υπάρχει και άλλος περιορισμός θα έλεγα που είναι η αξιολόγηση που κάνει η Επιτροπή των δράσεων και προγραμμάτων αυτών. Για το ένα β κοινωνικό ταμείο 1,9% δεσμεύσεις. Η συνολική βεβαίως αύξηση έχει ως στόχο να μειώσει τα μη καταβληθέντα, όπως έλεγα και νωρίτερα. Το Ταμείο Ενίσχυσης των Απόρων αυξάνει κατά 2% και τελικά 26,9 για τις πραγματικές καταβολές και συγκρίνουν το 15. Για την πρωτοβουλία για τους νέους, για την απασχόληση και το είχα γράψει στην έκθεση της εντολής ίσως έχουμε κάποιους συναδέλφους που δεν έχουν αντιληφθεί ακόμα. Είχαμε κάνει το front loading της πρωτοβουλίας. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι το 16 δεν έχουμε πιστώσεις. Δηλαδή δεν έχουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε το μηχανισμό της πρωτοβουλίας. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσουμε και θα ήταν κακό σημάδι, σινιάλο υπό τις συνθήκες πολύ αυξημένης ανεργίας μεταξύ των νέων, να πούμε εμείς τελικά ότι ολοκληρώνουμε αυτό το πρόγραμμα, το πρόγραμμα που θα ήταν μόνο για 14-15, ενώ το 16 δεν έχουμε πλέον ποσά. Προτείνω λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε την ευελιξία για να υπάρξουν κονδύλια για τις πρωτοβουλίες. Τώρα θα μου πει κανεί υπάρχουν τόσα πολλά μη καταβληθέντα, μη χρησιμοποιηθέντα. Αυτό πρέπει να το δούμε. Πρέπει να ξαναδούμε κάποιους κανόνες, πρέπει να ξαναδούμε γιατί έχουμε τα φαινόμενα αυτά, γιατί δεν λειτουργούν τα πράγματα όπως θέλουμε. Πρέπει να δούμε επίσης τα κονδύλια των επιχειρησιακών προγραμμάτων που έχουν υιοθετηθεί. Αλλά ε, βεβαίως για μένα είναι θέμα προτεραιότητας το θέμα της ενεργείας των νέων. Πρέπει πρώτα να χρησιμοποιήσουμε τα ποσά που έχουμε διαθέσιμα, τα εξειδείς που κάναμε front loading, αλλά και να χρησιμοποιήσουμε με το πρόγραμμα αυτό και επ' αυτού υιοθετώ και τη θέση αυτή που σας περιγράφω και ελπίζω να έχω τη στήριξη των μελών γιατί νομίζω πραγματικά ότι πρέπει να συνεχιστεί αυτή η πρωτοβουλία. Νομίζω ότι τα πιο σημαντικά τα ανέφερα. Αναφέρθηκα και στις πληρωμές. Άρα σας ακούω για να έχουμε τον καλύτερο δυνατό προϋπολογισμό με τους περιορισμούς που ξέρουμε ότι έχουμε. Έγινε το σχέδιο προϋπολογισμού από την Κομισιόν, το Συμβούλιο θα κάνει τη δική του ανάγνωση, τα μεγέθη που σας ανέφερα θα διαβαστούν και θα ερμηνευθούν από το Συμβούλιο και θα δούμε πώς θα τα ερμηνεύσει το Συμβούλιο. Ξέρουμε ότι πάντα προσπαθεί να περιορίσει ακόμα περαιτέρω έναν ήδη περιορισμένο προϋπολογισμό από το Συμβούλιο. Προσπαθεί να μειώσει σε σχέση με τη χρήση των περιθωρίων, σε σχέση με τη χρήση των κονδυλίων που ήδη είναι ανεπαρκή, θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Εγώ θα ήλπιζα, θα ήλπιζα, θα ευχόμουν το Συμβούλιο να τηρήσει τις δεσμεύσεις και υποσχέσεις που ανελήφθησαν ε, ή στα πλαίσια του πολιετού δημοσιονομικού, αλλά και σε σχέση με τις διακηρύξεις και ανακοινώσεις του Συμβουλίου οι οποίες όμως ποτέ δεν βρίσκουν το δρόμο τους προς αυτά χρηματοδοτικά μέσα. Σας ευχαριστώ. Thank you, Mr. Ευχαριστώ κύριε Φερνάντες. Ξέρετε ότι στις 9.30 ψηφίζουμε. Δεν θα ξεκινήσουμε 9.30 γιατί πρέπει να ακούσουμε κάποια σχόλια γύρω από αυτό. Αλλά παρακαλώ να είσαστε πάρα πολύ σύντομοι. Θα δώσω το λόγο στον εισηγητή, στην εισηγήτρια, την κυρία Κλιούν. Και πέραν αυτού έχω τους κυρίους Μπάλας, Μωρέν Σαρτιέ, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος άλλος, Ριμπέιρο. Μετά επιστρέφουμε στον κύριο Φερνάντες και να αρχίσουμε τις ψηφοφορίες. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Κλούν. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Φερνάντες για την παρουσία σας εδώ σήμερα. Εμείς θα συζητήσαμε τα θέματα αυτά στις πολιτικές ομάδες και στη δική μου και νομίζω καταλήξαμε σε συμβιβασμούς οι οποίοι καλύπτουν την πλειοψηφία. Εμείς θέλουμε πραγματικά να υπάρχει μια ισχυρή άποψη από πλευρά της Επιτροπής μας Αναφερθήκατε κι εσείς ο ίδιος κύριε Φερνάντε τα θέματα των νεότητας, του Ταμείου για την Νεότητα κτλ. Και το θέμα της ανεργίας των νέων είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί ιδιαίτερα, ιδιαίτερα αυτή τη δύσκολη εποχή. Έχουμε 22% μεσόρο ανεργίας των νέων με ιδιαίτερα υψηλά κορυφαία ποσοστά για ορισμένες χώρες. Παρατήρησα επίσης αυτά τα οποία είπατε και για το λεγόμενο front loading. Έχουμε συζητήσει τα θέματα αυτά μαζί με την κυρία Μωρέν Σαρτιέ στο παρελθόν. Πάντως, από τα σχόλιά σας καταλαβαίνω ότι και εσείς εμένετε στην πρωτοβουλία αυτή την οποία βρίσκουμε καθοριστική και θα πρέπει στα πλαίσια της αναζήτησης της ευελιξίας να ολοκληρώσουμε όλα τα προγράμματα γύρω από τους νέους. Είναι θέμα απόκτησης ικανοτήτων, είναι θέμα εκ νέου κατάρτισης, εκπαίδευσης στα της πράσινης οικονομίας. Αναφερθήκατε επίσης και στα τρία ή αγγλικό δηλαδή επιχειρήσεις, επιχειρηματικό πνεύμα, μικρομεσαίες, είναι ζωτικά παιδεία αυτά για τη δημιουργία θέσεων εργασίας πρέπει να βοηθήσουμε τις μικρομεσαίες είναι το κλειδί για τη δημιουργία των θέσεων αυτών. Ένα άλλο θέμα είναι το της μικροχρηματοδότησης και της διεύρυνσης της εμβέλειάς της. Λοιπόν, θέλω να πω ότι με λίγα λόγια μέχρι τώρα εμείς ε, έχουμε διαμορφώσει μια πρώτη γνωμοδότηση. Θα το συζητήσουμε το θέμα αυτό μπαίνοντα σε λεπτομέρειες σε σχέση με τα ποσά και με τους τρόπους χρηματοδότησης. Νομίζω ότι θα πρέπει να εμείνουμε κυρίως στην ανεργία των νέων, την υποστήριξη των μικρομεσαίων και την ανάκτηση επαγγελματικών ικανοτήτων και εκ νέου κατάρτιση για τους εργαζόμενους. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Μπάλας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα μιλήσω εξ ονόματος της Σοσιαλιστικής Ομάδας και του συναδέλφου Πυρίνσκι το θέμα του προϋπολογισμού είναι ένα περίπλοκο θέμα και έχουμε μπροστά μας όργανα που ονειρεύονται να μειώσουν ακόμα περισσότερο την προσπάθεια την οποία εμείς κάναμε. Πρέπει λοιπόν να αποκαταστήσουμε μια κάποια ισορροπία. Εξ αυτού αυτά τα οποία μας περιμένουν στο κοινωνικό ταμείο είναι προβληματικά ή και εμβληματικά της κατάστασης η οποία επικρατεί. Τα χρήματα δεν χρησιμοποιούνται με σωστό τρόπο από, ορισμένους, από ορισμένες χώρες και βρισκόμαστε πλέον σε μια κατάσταση όπου είμαστε υποχρεωμένοι να δεχθούμε κάποιες ε, εκ των ρυθμίσεις του προϋπολογισμού. Δηλαδή ενώ υπάρχουν ανάγκες δεν χρησιμοποιούμε όλες τις διαθέσιμες πιστώσεις για να μειώσουμε τον προϋπολογισμό. Βλέπουμε λοιπόν ότι εκεί έχουμε κάποιο πρόβλημα. Για το ΑΒ, το ΑΑ έχουμε ε, ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε σχέση με την Ευρώπη 2020 ε, ε, εμείς να στηρίξουμε νέους πόρους για τον προϋπολογισμό, ισχυρούς πόρους για τον προϋπολογισμό, όσο πιο απομεμακρυσμένους από τα κράτη γίνεται. Ξέρω ότι είναι μια ουτοπία αυτή, αλλά πρέπει να παίξουμε πάνω σε αυτό για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε αυτόνομα από τα κράτη-μέλη. Θα πρέπει λοιπόν να στηρίξουμε την προσπάθεια αυτή η οποία γίνεται αλλά όντας ιδιαίτερος προσεκτική και σε σχέση με τους πόρους και σε σχέση με τη συγκεκριμένη χρήση των πόρων αυτών που δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί εκ των υστέρων για μείωση περαιτέρω δημοσιονομική. Ευχαριστώ πολύ. Euh, να ευχαριστήσω τον κύριο Φερνάντες που μας παρουσίασε την εργασία του σήμερα το πρωί. Πρέπει να είμαστε σε τέσσερα σημεία πολύ επιφυλακτικοί. Το πρώτο είναι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και ό,τι έχει σχέση με την πολιτική της απασχόλησης. Στα πλαίσια του κοινωνικού ταμείου, όπως είπατε με κάθε ειλικρίνεια, υπήρξαν τόσα υπόλοιπα και τόσοι μη πληρωμένοι λογαριασμοί, στην ουσία βλέπουμε ότι μειώνουμε τους πόρους ε, της ε, φετινής χρονιάς, γιατί ε, τα χρησιμοποιούμε τα χρήματα αυτά για να καλύψουμε τις περσινές τρύπες. Κοιτάξτε, δεν πληρώσαμε αυτό που έπρεπε να πληρώσουμε. Και εδώ οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων θα πρέπει ε, να μην πιστεύουν ότι με τέτοια μέτρα θα προωθήσουν την πολιτική της απασχόλησης. Δυστυχώς το μόνο που κάνουμε είναι να βουλώνουμε τις περσινές τρύπες. Δεύτερο θέμα είναι η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων στην οποία επιμείνατε. Το κύριο πρόβλημα το οποίο εγώ διακρίνω είναι ότι μόλις ψηφίσαμε εδώ τον μήνα Απρίλιο, αν δεν κάνω λάθος, το θέμα της προχρηματοδότησης κατά 30% για την πρωτοβουλία για τους νέους, για να δώσουμε κίνητρα. Και το κάναμε σε χρόνο ρεκόρ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μέσα σε ένα τρίμηνο, Επιτροπή και εμείς καλύψαμε προχρηματοδότηση 30% για την πρωτοβουλία για τους νέους. Και τώρα θα βρεθούμε με μια τρύπα στον προϋπολογισμό. Δεν είναι δυνατόν. Πρέπει να διασφαλίσουμε τη συνέχεια ανάμεσα στις πολιτικές δράσεις τις οποίες έχουμε αναλάβει και τον προϋπολογισμό που δεν είναι παρά η μετάφραση σε δημοσιονομικούς όρους της πολιτικής μας επιλογής. Τρίτο θέμα είναι το Ταμείο για την Παγκοσμιοποίηση. Εμείς για αυτό το Ταμείο τόσα χρόνια δουλεύουμε, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων στην ουσία μειώνουν τη χρηματοδότηση αλλά αυξάνονται από τα κράτη-μέλη βέβαια οι αιτήσει για χρηματοδότηση. Έχουν ανάγκη από αυτό το ταμείο και τα χρήματα αυτά δεν πηγαίνουν σε επιχειρήσεις, πηγαίνουν σε εργαζομένους για να μπορέσουν να κάνουν μια νέα επαγγελματική εκπαίδευση. Δεν μπορούμε λοιπόν εδώ να σφυρίζουμε κλέφτικα. Δεν πρέπει να υποχωρήσουμε ούτε φυσικά. Και στο τέλος τώρα για το Ταμείο, για, τους, ε, για την ακραία φτώχεια κτλ. Ε, εμείς σώσαμε την πρόταση που είχε γίνει παρά την προσπάθεια του Συμβουλίου. Πρόκειται για το σημείο το οποίο ενδιαφέρει περισσότερο αν θέλετε τα μέσα ενημέρωσης και την κοινή γνώμη. Εάν η Ευρώπη δεν είναι σε θέση να αναλάβει τη συγκεκριμένη υποχρέωση και να τη φέρει εις πέρας, τότε η εικόνα που θα δώσουμε θα είναι απαράδεκτη. Ευχαριστώ κυρία Ριμπέιρο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον κύριο Φερνάντες που ήρθε σήμερα εδώ για να συζητήσει μαζί μας. Δύο βασικά στοιχεία από αυτά που αναφέρατε θα ήθελα να σχολιάσω. Καταρχάς, την ανάγκη να επενδύσουμε και να βοηθήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μας καθώς και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις μας να επενδύσουν. Και επίσης θα ήθελα να σχολιάσω τις κοινωνικές πολιτικές όσον αφορά την νεολαία και την απασχόληση. Ο Σωσέ Μανουέλ αναφέρθηκε στα νέα προγράμματα από το 2016. Θα πρέπει να υπάρχει συνέχεια ανάμεσα στα διάφορα προγράμματα, αλλά αυτή διακυβεύεται αυτή τη στιγμή. Πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιηθούν οι πόροι από την εγγύηση για την νεολαία. Και όσον αφορά την ευελιξία, που είναι κάτι το οποίο υπερασπιστήκατε, όσον αφορά το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, θα ήθελα να ρωτήσω, υπάρχουν στοιχεία σχετικά με τα μη απορροφημένα ποσά των τελευταίων ετών στα διάφορα κράτη-μέλη και ποια είναι η θέση της Επιτροπής σε σχέση με την ευελιξία αυτή. Ευχαριστώ. Ε, θα δώσω το λόγο στον κύριο Φερνάντη για να κλείσει τη συζήτηση. Ε, να ευχαριστήσω και εγώ ε, για τα σχόλιά σας. Για τον προϋπολογισμό είναι σαφές ότι ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι κάτι το οποίο αρκεί. Είναι μικρός, αλλά παρότι είναι μικρός είναι πολύ σημαντικός και σε κάποιες χώρες αντιπροσωπεύει άνω του 50% των επενδύσεων. Υπάρχει επίσης κάτι το οποίο θα πρέπει να επαναλαμβάνουμε συνεχώς. Ο προϋπολογισμός μας είναι επενδυτικός, 94%. Αυτό σημαίνει ότι μόνο το 6% είναι οι λειτουργικές δαπάνες και οι διοικητικές δαπάνες. Αυτό αποδεικνύει την προστιθέμενη αξία του προϋπολογισμού αυτού. Έχει ένα πρόβλημα βέβαια, αλλά δεν θα το συζητήσουμε σήμερα γιατί θα θέλαμε πάρα πολύ χρόνο, ότι δηλαδή το 85% των εσόδων προέρχονται από, τα εθνικ, από εθνικούς πόρους και έχουμε ανάγκη από ιδίους πόρους, από πραγματικούς ιδίους πόρους. Συμφωνώ για τις προτεραιότητες, το είπα και εγώ, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό ταμείο. Και τα άλλα ταμεία της συνοχής είναι επίσης σημαντικά για την απασχόληση. Ακόμα και το σχέδιο επενδύσεων, στρατηγικό σχέδιο ε, του Ιούνκερ έχει μεγάλο ρόλο να παίξει στον τομέα της απασχόλησης. Θα πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε και να σεβαστούμε ε, τις συμβιβαστικές ε, προτάσεις. Το είπα αυτό εξ αρχής. Αν δούμε το πολιετές δημοσιονομικό 14-15 ναι, είναι αλήθεια ότι στην ουσία καλύπτουμε το παρελθόν, τα κενά του παρελθόντος. Το πραγματικό, το ουσιαστικό νέο δημοσιονομικό θα ξεκινήσει από του χρόνου ουσιαστικά. Αυτό σημαίνει ότι οι συμβιβαστικές προτάσεις ε, ε, δεν καλύπτουν απόλυτα τον πλήρη σεβασμό του, πολυ, του πολιετούς. Τώρα, η πρωτοβουλία για τους νέους. Δεν έχω ακριβώς όλα τα στοιχεία που χρειάζεται θα τα συλλέξω και θα σας απαντήσω για το θέμα της εκτέλεσης που είναι πολύ σημαντικό. Να μην ξεχνάμε ότι έχουν υπάρξει πολλές καθυστερήσεις στα λειτουργικά προγράμματα. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν καθυστερήσεις για την θέση σε λειτουργία αυτής της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων. Έχω ξεκινήσει λοιπόν και χαίρομαι γιατί συμφωνείτε έτσι ώστε από το 2016 να υπάρξουν συγκεκριμένες πιστώσεις υποχρεώσεων που θα διασφαλίζουν τη συνέχεια της πρωτοβουλίας αυτής. Θα πρέπει να σταματήσουμε λοιπόν να τελειώνουμε με τα υπόλοιπα από το παρελθόν το 2016. Βέβαια αυτό το οποίο συμβαίνει το 2014-2015... Έχουμε τρία χρόνια, είναι ο κανόνας νήσιν τρία, εδώ μην το ξεχνάμε. Είμαστε στο εσωτερικό του ε, κοινωνικού ταμείου, αλλά από την άλλη το 2016 δεν θα καταλάβει ο κόσμος αν δεν υπάρξουν νέες πρωτοβουλίες για τους νέους. Τώρα για το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης νομίζω ότι 30 δις πληρωμές ε, είναι κάτι το οποίο είναι λίγο. Γενικά ε, θα πρέπει να δούμε ε, ποιοι είναι αυτοί που χρησιμοποιούν περισσότερο το ταμείο αυτό και ταυτόχρονα διαμαρτύρονται για τις αυξήσεις του. Λοιπόν, Έχουμε κάποια περιθώρια. Είχαμε για το 2015 ε, ένα δις 500 περίπου εκατομμύρια. Θα χρησιμοποιήσουμε ένα τμήμα όμως για ε, το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Το 2016 το περιθώριο είναι 2,2 δις. Θα πρέπει επίσης να υπενθυμίσουμε ότι το 1,1 δις είναι στον τίτλο 2, δηλαδή έχουμε ένα περιθώριο άνετο σχετικά, αλλά έχουμε και επίσης κάποια επιπλέον μέσα ευελιξίας. Όταν μιλάμε για το Ταμείο Παγκοσμιοποιήσεως πρόκειται για ένα ειδικού τύπου μέσο. Υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις στις θέσεις μας με το Συμβούλιο για αυτά τα ειδικά μέσα. Εμείς θεωρούμε ότι τα ειδικά μέσα είναι εκτός προϋπολογισμού και εκτός πολιετούς δημοσιονομικού. Δεν συμπεριλαμβάνονται στον γενικό λογαριασμό. Έχουμε την δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα μέσα ευελιξίας λοιπόν έτσι ώστε να καλύψουμε την ανάγκη που δημιουργείται για την απασχόληση των νέων και στις υποχρεώσεις αλλά είπα ότι το 16 θα υπάρξει κάτι το εντελώς νέο το οποίο είναι το λεγόμενο γενικής φύσης περιθώριο που δεν είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Τα χρήματα τα οποία δεν χρησιμοποιούνται τότε πηγαίνουν σε ένα γενικό περιθώριο και τότε μόνο μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για πολιτικούς στόχους, ιδιαίτερα την απασχόληση και την ανάπτυξη. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Το έχω υπενθυμίσει επανειλημμένα στις διαπραγματεύσεις για το σχέδιο Juncker. Το Συμβούλιο θέλει να το ξεχνάει αυτό. Το Συμβούλιο εξακολουθεί ε, να εργάζεται σύμφωνα με το προηγούμενο δημοσιονομικό πλαίσιο. Το άρθρο 14 του πολιετούς πλαισίου λέει ότι τα περιθώρια των μη χρησιμοποιούμενων υποχρεώσεων πηγαίνουν σε ένα νέο περιθώριο σφαιρικό, συνολικό, γενικής φύσεως που μπορεί να χρησιμοποιείται για πολιτικούς στόχους όπως η ανάπτυξη και η απασχόληση. Και μάλιστα λέγεται εκεί για την απασχόληση των νέων, για την προώθηση της απασχόλησης των νέων. Βλέπετε λοιπόν ότι μιας και έχουμε αυτά τα στοιχεία στον προϋπολογισμό ε, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον ε, συμβιβασμό αυτό του Συμβουλίου. Νομίζω ότι οι διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο επί του Δημοσιονομικού είναι πάντα δύσκολες στην αλήθεια, αλλά θα κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι ώστε να υπάρξει σεβασμός των συμβιβασμών αυτών. Ε, γιατί είναι ντροπή η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί ε, έχουμε πει ότι πάκτα sunt servanda», τα υπεσχημένα τηρούνται. Λοιπόν, στη συγκεκριμένη περίπτωση διαπιστώνουμε, είναι ντροπή να πληρώνουμε επιτόκια λόγω της καθυστέρησης στις πληρωμές. Οι πληρωμές που είναι συνέπεια λογική απλά των υποχρεώσεων τις οποίες έχουμε υιοθετήσει. Δεν θα έπρεπε να το συζητάμε, θα έπρεπε να πληρώνουμε γιατί όταν πληρώνουμε τότε αναφερόμαστε σε αυτά τα οποία έχουν ήδη σημειωθεί για συγκεκριμένη χρήση, για μικρομεσές για τις απόμακρες περιφέρειες, για τις τοπικές αρχές, για την απασχόληση των νέων. Πρόκειται για χρήματα τα οποία έχουν ουσιαστικά ήδη δαπανηθεί. Σας ευχαριστώ και υπολογίζω στην υποστήριξή σας. Ελπίζω να καταλήξουμε γρήγορα. Thank you, Mr. Fernandez, for your strong Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις θέσεις που μας παρουσιάσατε και θα σας υποστηρίξουμε στον αγώνα σας ε, να διατεθούν πολλά χρήματα για την καταπολέμηση της ανεργίας. Σας ευχαριστώ που ήρθατε εδώ. 22 με 23 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η ψηφοφορία στην Επιτροπή Προϋπολογισμού και θα πάει στην Ολομέλεια του Ιουλίου. Σε δύο-τρία λεπτά θα ξεκινήσουμε τις ψηφοφορίες. Okay, then we'll start with the voting. Ξεκινήσουμε τις ψηφοφορίες λοιπόν. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Παγκοσμιοποίησης για την περίπτωση Broadcom από τη Φιλανδία. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Ποιος είναι υπέρ, παρακαλώ. Λήξη της ψηφοφορίας. Ευχαριστώ πολύ. Περνάμε στις κατευθυντήριες ε, γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησεις των κρατών μελών. Τροπολογία 101. Ποιος είναι υπέρ. Ποιος είναι κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική και η κάπα. Ποιο είναι υπέρ, κατά, απόχέ εγκρίνεται. Συμβιβαστική L. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική M. Μη. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 127 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική ΑΒ υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 129 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 130 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική νη υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική NA υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 141 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 142 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική όμικρον υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 151 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική π υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 157 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική Q υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Θα ελέγξουμε την 157 λέει η Πρόεδρος. Όχι. Την συμβιβαστική Q. Αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 28 ψήφοι υπέρ. Τροπολογία 170, 170 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική ρο υπέρ Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 177 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική S υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική T ταφ υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική U υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 189 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά την τροπολογία 189 αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας εγκρίνεται με 24 ψήφους υπέρ. Συμβιβαστική Β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική W υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 212 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 213. 213 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 214 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική Y, Y, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική ζήτα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική ΑΑ υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 245 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 246 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 34 υπέρ κατά αποχές να την ελέγξουμε. Uh, the vote is closed and is carried by 29 votes. Λήξη της ψηφοφορίας εγκρίνεται με 29 ψήφους. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ελέγχουμε την τροπολογία 3. Αρχή της ψηφοφορίας. the vote is closed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 Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 56. Ψηφοφορία κατά θύματα. Το πρώτο μέρος υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Το δεύτερο μέρος υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Να ελέγξουμε το δεύτερο μέρος της τροπολογίας 56. The Αρχή της ψηφοφορίας, λήξη της ψηφοφορίας. And it is rejected. Απορρίπτεται. Τροπολογία 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 57. Καταπίπτει. Όπως και η 58. Συμβαστική C υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Compromise D. Συμβιβαστική D υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Να ελέγξουμε τη συμβιβαστική D, αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Compromise E, those in favor. Συμβιβαστική ε, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 67 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 68 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται να ελέγξουμε την 68 αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 22 ψήφοι υπέρ. Συμβαστική F. Με προφορική τροπολογία του ΕΛΚ. Problem? Are there objections to the oral There are objections to the other amendment. Mm, okay. Uh-huh. So we vote on the original text. There are objections. We stick to the original text uh, uh, and. Uh, uh, Υπάρχει αντίρρηση, οπότε θα εμείνουμε στην αρχική διατύπωση. Συμβαστική F υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική G υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική H υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική Ι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 94 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 96 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική J υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Θα ψηφίσουμε το σύνολο της έκθεσης όπως τροποποιήθηκε. Αρχή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. εγκρίνεται με 37 ψήφους υπέρ και 6 ψήφους κατά. Ευχαριστώ την κυρία Άγκαια. Και προχωράμε. the Green Initiative and we start with Πρωτοβουλία για την πράσινη απασχόληση, συμβαστική J, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 53, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 55 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Να ελέγξουμε την τροπολογία 55. Ψηφίζετε παρακαλώ. Λήξη της ψηφοφορίας απορρίπτεται. Εκτός μικροφώνου παρατηρήσεις δεν ακούμε. Μπορούμε να συνεχίσουμε. Ωραία. Προχωράμε στην NV2, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. NV3, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. NV5 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. NV6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική L υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 61 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. ΦΕΜ 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται θα έλεγα. Να ελέγξουμε. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβαστική M, μη, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική N, νη, υπέρ, κατά, Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 64 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 65 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 66 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική όμικρον υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 76 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Θα ελέγξουμε την τροπολογία 76 ηλεκτρονικά. Παραμένει ανοιχτή η ψηφοφορία. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Κατά μία ψήφο. 77 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική Q υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. «83 υπέρ». «Κατά αποχές εγκρίνεται». 84 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική R, ρο, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 87 θα γίνει ψηφοφορία κατά τμήματα. Το πρώτο μέρος υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο μέρος υπέρ, κατά, να την ελέγξουμε. Ελέγχουμε λοιπόν το δεύτερο μέρος της τροπολογίας 87. Αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με 27 ψήφους υπέρ. Συμβαστική S. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 91 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Να ελέγξουμε την 91 υπέρ. Ε, συγγνώμη, αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται κατά δύο ψήφους. 93 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 94 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική T υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική TA υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. ΦΕΜ 3 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ελέγχουμε την ΦΕΜ 3. And the vote is now closed. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται κατά τέσσερις ψήφους. ΦΕΜ 4 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 99 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 100 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 101 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 102 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική U υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική V υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την τροπολογία 106 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Θα ελέγξουμε την 106. λήξη της ψηφοφορίας ε, εγκρίνεται κατά τρεις ψήφους. Φέμε 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 110 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική W υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 116 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεν ήταν η τελευταία τροπολογία. Τροπολογία 117 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική XA υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ελέγχουμε τη συμβαστική XA. The Λήξη της ψηφοφορίας απορρίπτεται. ΦΕΜ 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Φεμ 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Φεμ 14 υπέρ Καταπίπτει. Όχι, όχι, δεν καταπίπτει. Φεμ 14 υπέρ κατά αποχές πρέπει να την ελέγξουμε. Φεμ 14 αρχή της ψηφοφορίας. And uh, now it's closed. And it's uh, rejected. Λήξη της ψηφοφορίας απορρίπτεται. Κατά 6 ψήφους. ΦΕΜ 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. ΦΕΜ 13 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. ΦΕΜ 17 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική Y, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 123 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική Z, Z, υπέρ, κατά αποχές. Αν δεν είδα καλά πρέπει να το ελέγξουμε. Συμβαστική Z. Αρχή της ψηφοφορίας λήξη της ψηφοφορίας εγκρίνεται με 40 ψήφους. Δεν σκόσατε τα χέρια σας όμως. 24 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 130 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 131 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται να ελέγξουμε την 131 αρχή της ψηφοφορίας. Still open. Okay. Then we close the votes. Yes. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται κατά πέντε ψήφους. 132 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική ΑΑ υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική ΑΒ υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική AC υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. NV29 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 140 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική AD υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 147 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 148 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 149 υπέρ κατά αποχές Ίσως να μπορείτε, δεν είμαι βέβαιη. Ελέγχουμε λοιπόν την 149. Λήξη της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Συμβαστική ΑΕ υπέρ κατά αποχε εγκρίνεται. Συμβαστική ΑΕΦ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. NV19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. NV20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε μαζί τις τροπολογίες 153, 154, 155 και 156. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Να ελέγξουμε. Αρχή της ψηφοφορίας. 153 έως 156 είναι οι τροπολογίες που ψηφίζουμε. Λήξη της ψηφοφορίας απορρίπτονται. 157 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 158 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 159 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 160 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική AFA υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται θα έλεγα. πρέπει να ψηφίσουμε την NV21. Υπάρχει λάθος στον κατάλογο της ψηφοφορίας. Πρέπει λοιπόν να ψηφίσουμε την NV21 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. NV22 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 162 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβεβαστική AG, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Να δω ένα λεπτό. 168 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να την ελέγξουμε. The and the vote is open. Άρχεται η ψηφοφορία στην 168 πέρας της ψηφοφορίας απερίφθη κατά 10 NV23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 169 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται M25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 170 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 172 υπέρ κατά αποχές MV26 υπέρ κατά αποχές MV27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται MV28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική AH υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και πάμε απευθείας στην συμβιβαστική ΑΙ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. AG λέει η πρόεδρος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ε, 188 those in favor those... 188 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 189 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 190 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 191 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Φεμ 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 192 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 193 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 194 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική κάπα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 196 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική AL υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται NV11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται NV12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται MV13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 198 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 199 υπέρ κατά αποχές να την ελέγξουμε την 199 άρχεται η ψηφοφορία Όχι, το συγγνώμη, λέει ο πρόεδρο. Υπήρξε ισχυρότατη στήριξη. Λοιπόν, ΦΕΜ 11, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. 200 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 201 ε, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. NV34 καταπίπτει, όχι. Είναι, είναι ακόμα εκεί, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. NV35 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. NV36 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 202 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 203 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 204 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται όχι να την ελέγξουμε το 204 είναι ακόμα ανοιχτή η ψηφοφορία λέει ο πρόεδρος και τώρα κλείνει και απορρίπτεται. 205 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Όχι να ελέγξουμε. Να ελέγξουμε 205. Πέρας τις ψηφοφορίες απορρίπτεται κατά τέσσερις ψήφους. 206 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 207 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 208 υπέρ κατά από την αρχή 208 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται λέει η πρόεδρος. Όχι, ελέγχουμε τη 208. And the vote is... Πέρα στις πληροφορίες. Ναι, απορρίπτεται. Κατά μία ψήφο. Συμβαστική α, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική σε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική Δ. υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 48 υπέρ κατά απόχες εγκρίνεται. Συμβαστική ε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική F υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική G υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 34 υπέρ κατά αποχές ίσως και να εγκρίνεται να την ελέγξουμε την 34 πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται κατά 33 ψήφους 35 υπέρ κατά Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική H υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική γιώτα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 46 υπέρ το πρώτο τμήμα της 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα της 46 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Να ελέγξουμε την, το δεύτερο τμήμα της 46. Ψηφίζομαι και πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται με τρεις ψήφους. Λοιπόν, 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Φεμ H υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. έλεγχος, έλεγχος στην Φεμ H. Πες, ε, ε, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται κατά πέντε ψήφους. Φεμ J υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ελέγχουμε την Φεμ Άρα άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται κατά πέντε. 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 51 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και πάμε στην 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και ψηφίζουμε στην ούτως τροποποιημένη έκθεση με ηλεκτρονική ψηφοφορία άρχεται η ψηφοφορία ονομαστική εγκρίνεται κατά 41 ψήφους. Συγχαρητήρια. we'll the... Πάμε τώρα στο σχέδιο γνωμοδότησης του προϋπολογισμού για το 16. Συμβαστική α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τρία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τρία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίας. Απερίφθη η τρία. Δεν το κατάλαβα εγώ. Περνάμε στην 7 τώρα. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος τότε για την 7. Πέρα στις ψηφοφορίες δεκτή 28 υπέρ. Συνεχίζουμε στην 1β μικρό τροπολογία 8 ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. Συμβιβαστική β κεφαλαίο υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Δεκαπέντε υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. Συμβιβαστική γάμα υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 20 υπέρ, κατά, αποχές, αποχές, απερίφη. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 20 παρακαλώ. Δεν έχει κλείσει ακόμα η ψηφοφορία. Τώρα απερίφθη με δύο ψήφους διαφορά. 21 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. D υπέρ κατά αποχές δεκτή. 25 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 27 υπέρ κατά αποχές απερίφη 28 υπέρ κατά αποχές απερίφη 28 ελέγχουμε άρχεται η ψηφοφορία πέρας της ψηφοφορίας Γίνεται δεκτή με 8 ψήφους διαφορά. 29 ψηφίζουμε. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη 29. Ψηφίζουμε την 30 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 31 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. Συμβιβαστική ή αγγλικό υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 35 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 36 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 37 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Η 38 απεσήφθη. Η 39 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 40 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 41 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. Συμβιβαστική F. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 47 ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Συμβιβαστική G ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 53 ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 54 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 55 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 56 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Σύνολο τροπολογημένη νομοδότηση ονομαστική ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας Σαράντα υπέρ κατά γίνεται δεκτή. Σας ευχαριστώ όλους. Το επόμενο θέμα τώρα στην ημερήσια διάταξη Πάμε αρκετά πιο γρήγορα. Έξι λεπτά πιο γρήγορα. Πάμε λοιπόν στο 11. Εξουσιοδότηση των κρατών μελών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 Okay, we start uh, with point 11 on the agenda uh, Ξεκινάμε με το 11. Αδειοδότηση λοιπόν, εξουσιοδότηση των κρατών μελών για κύρωση πρωτοκόλλου του 2014 για τη Σύμβαση για Αναγκαστική Εργασία της ΔΟΕ σχετικά με θέματα που αφορούν την κοινωνική πολιτική. Ζητείτε εμείς να συμφωνήσουμε με την προτινόμενη πράξη, δηλαδή την πρόταση του Συμβουλίου επί τη βάση ακριβώς της Επιτροπής Απασχόλησης. Είναι αρκετά σημαντικό θέμα λοιπόν και θα δώσω το λόγο στον Πατρίκ Λεοιαρίκ από την ΚΟΕ. Έχετε το λόγο κύριε Λεοιαρίκ. Παρακαλώ όσοι βγαίνετε από την αίθουσα να κάνετε ησυχία. Ο κύριος Λουιαρικ. Πρόεδρε, συνάδελφοι, μιλάμε για την επικύρωση του πρωτοκόλου του 2014 της Διεθνούς Οργάνωσης για την Εργασία για την επικαιροποίηση της Σύμβασης για την Αναγκαστική Εργασία η οποία ισχύει από το 1930 εκπλήσει η τόσο καθυστερημένη επικαιροποίηση. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της ΔΟΕ, η αναγκαστική υποχρεωτική εργασία δυστυχώς αφορά 21 εκατομμύρια ανθρώπους στον κόσμο. Οπότε οι αλλαγές αυτές είναι καλές. Από τις Φιλιππινέζες υπηρέτριες, τις οποίες εκμεταλλεύονται στην Ευρώπη, από αυτούς που εκμεταλλεύονται όσους περνούν παράνομα τα σύνορα, όσοι εργάζονται στην κατασκευή των γηπέδων του Κατάρ ή σε αυτούς που εκμεταλλεύονται τις γυναίκες και τα παιδιά για σεξουαλικούς λόγους οι πολίτες σε αυτόν τον κόσμο υποφέρουν. 150 δις κατέτος για όσους οργανώνουν τέτοιες μορφές εργασίας. Αυτό δεν μπορούμε λοιπόν να το δεχτούμε πλέον. Στις παραδοσιακές μορφές εκμετάλλευσης προστίθενται και νέες μορφές στις πλούσιες χώρες παρά την ύπαρξη του κράτους δικαίου. Πιο ύποπτες, πιο διακριτικές, πιο υπόγειες αλλά εξίσου βίες είναι οι μορφές εκμετάλλευσης της ελπίδας για μια καλύτερη ζωή όλοι οι άνδρες, όλες οι γυναίκες, όλα τα παιδιά που θέλησαν να φύγουν από τις χώρες τους και να έρθουν παράνομα στην Ευρώπη με δραματικές συνθήκες. Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας είναι 1,5 εκατομμύριο περίπου στο σύνολο της Υπήρου μεταξύ των οποίων ένα μεγάλο τμήμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που υποφέρουν από την υποχρεωτική εργασία, άνθρωποι στους οποίους υποσχεθήκαμε μια δουλειά στο εξωτερικό, παγιδεύτηκαν λοιπόν ε, και πολλά παιδιά φυσικά υποφέρουν από την εκρίζωση την οποία υπέστησαν από τις χώρες τους. Οι πιο ευαίσθητες κατηγορίες του πληθυσμού, οι γυναίκες, τα παιδιά, οι μετανάστες είναι αυτοί που κάνουν τις χειρότερες δουλειές και κάτω από τις πιο απαράδεκτες συνθήκες, πορνεία, ζητιανιά και εδώ στην βία της εκμετάλλευσης προστίθεται και ψυχολογική βία και σωματική βία, φόβος και απομόνωση. Η απομόνωση αυτή η νέα μορφή σωματεμπορίας θα έλεγα πρέπει να απαγορευθούν μέσω νομικών ρυθμίσεων που θα γίνονται σεβαστές. 80 χρόνια μετά λοιπόν επικαιροποιείται η σύμβαση αυτή αποκτώντας νέα μέσα δράσης ε, εναντίον της κατανανταστικής εργασίας δίδοντας ένα δεσμευτικά νομικό χαρακτήρα. Το πλαίσιο και οι μορφές της υποχρεωτικής εργασίας έχουν πλέον αλλάξει και γι' αυτό το πρωτόκολλο όπως λέγει εδώ είναι απαραίτητο να ληφθούν μέτρα με τους κοινωνικούς εταίρους σε εθνικό επίπεδο και να καταπολεμηθεί το φαινόμενο. Το φαινόμενο αυτό περιλαμβάνει κάποιους συγκεκριμένους στόχους στο άρθρο 2, ενημέρωση των πληθυσμών που θεωρούνται ευάλωτοι, των εργοδοτών για να μην κρυθούν συνένοχοι, προστασία κυρίως των μεταναστών εργαζομένων, εφαρμογή του δικαίου της εργασίας, ενίσχυση των επιθεωρήσεων εργασίας, έλεγχος και του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Πολλά θα ήθελε να πει κανείς για τις βαθιές αιτίες αυτής της κατάστασης, την εκμετάλλευση των χωρών του Νότου από τις βόρειες χώρες, την ανισότητα των εμπορικών δικτύων, που οι νέες εμπορικές συμφωνίες δεν θα κάνουν τίποτα άλλο από το να χειροτερεύσουν. Η καταστροφή της αγροτικής γεωργίας κτλ. Επανέρχομαι στο πρωτόκολλο. Ένα από τα βασικά τμήματα είναι οι ευθύνε τις οποίες δίνει στα κράτη-μέλη στα άρθρα τα οποία καλύπτουν την υποχρέωση προστασίας των θυμάτων υποχρεωτικής εργασίας, την ευθύνη των κρατών μελών για μηχανισμούς αποζημίωσης και αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί διευκρινίζεται ανεξαρτήτως του καθεστώτος παραμονής του στο εθνικό έδαφος. Τέλος, ανάληψη υποχρέωσης έτσι ώστε καμία διαδικασία να μην αναλαμβάνεται εις βάρος των θυμάτων αυτής της καταναγκαστικής εργασίας. Και επίσης συνεργασία ανάμεσα στις συνυπογράφουσες χώρες για την αντιμετώπιση αυτής της αιώνιας θα έλεγε κανείς μορφής εκμετάλλευσης. Κάποιες χώρες όπως το Κατάρ ήταν κατά της επικύρωσης αυτού του πρωτοκόλου. Από τη δική μας πλευρά και μιας και μιλάμε για ευθύνες, θεωρούμε ότι είναι δική μας ευθύνη έτσι ώστε το πρωτόκολλο αυτό να επικυρωθεί το ταχύτερο δυνατόν. Η διαδικασία υιοθέτηση είναι μια διαδικασία απλοποιημένη η λεγόμενη της σύμφωνης γνώμης. Δηλαδή, εμείς δεν μπορούμε παρά να δώσουμε ή να αρνηθούμε τη σύμφωνη γνώμη μας. Κάτι το οποίο ε, αποκλείει τη διαδικασία τροπολόγησης. Εγώ λοιπόν υπόκειμαι στον κανόνα αυτό, ε, εξέφρασα γενικές σκέψεις, ε, δεν τροπολόγησα τίποτα. Εγκρίνοντας το πρωτόκολλο αυτό στην ουσία δημιουργούμε μια νέα διεθνή νομική πράξη μεγάλης εμβέλειας, ανθρωπιστικού χαρακτήρα. Η δεύτερη παρατήρηση την οποία θα ήθελα να κάνω είναι ότι το μέσον το οποίο επελέγει για την καταπολέμηση της εκμετάλλευσης αυτής είναι το δίκαιο μέσο της δημιουργίας και βελτίωσης του δικαίου εργασίας, δηλαδή του βασικού μέσου επί του οποίου βασίζεται το συγκεκριμένο πρωτόκολλο. Μου φαίνεται λοιπόν ότι είναι απαραίτητο για να υπενθυμίσουμε το νόημα αυτού του μέσου. Πρέπει λοιπόν να γίνει δεκτό το κείμενο αυτό το ταχύτερο δυνατόν. Θα πρέπει επίσης να συνεχίζουμε να υπερασπιζόμεθα το μέσο στο οποίο βασίζεται, δηλαδή το λεγόμενο θετικό δίκαιο εργασίας. Ευχαριστώ Πρόεδρε και συνάδελφοι για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ. Δίνω το λόγο στον κύριο Μπαχ που είναι σκιώδης εισηγητής από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Η αναγκαστική εργασία, όπως είπε ο εισηγητής, με όλες ε, τις συνέπειες που έχει για τους εμπλεκόμενους ε, αποτελεί ε, παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι άνθρωποι περιμένουν από εμά και από όλα τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφασιστική δράση ε, για να ε, αποτρέπεται η αναγκαστική εργασία και ελπίζουν σε εμάς και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό το ότι η ΔΟΕΣ ε, θέλει να συμπληρώσει την ε, σύμβαση με πρωτόκολλο του 2014. Υπόθηκαν πολλά, κάποια πράγματα ρυθμίζονται ήδη στην ε, κοινωνική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι όμως όλα και γι' αυτό είναι σημαντικό να δώσουμε στο Συμβούλιο την εξουσιοδότηση για επικύρωση όσο γίνεται πιο σύντομα ώστε να μπορέσει να ε, δράσει γρήγορα και προς όφελος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τις εργασίες του και θα ήθελα να εκφράσω την υποστήριξη του ΕΛΚ και ε, για την έκθεσή του και για την έκκληση προς τα κράτη-μέλη να επικυρώσουν όσο γίνεται πιο σύντομα το πρωτοκόλλο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Δίνω το λόγο στην Ιούτα Στάινρουκ, SND, που εκπροσωπεί τον σκιό Ευχαριστώ πολύ. Ο Μπράντο Μπενεφάη δεν μπορεί να είναι παρόν λόγω προβλημάτων με την πτήση του. Μπορώ όμως ε, εκ μέρους του να πω στον εισηγητή ότι τον ευχαριστεί για την δουλειά του και τον στηρίζει απολύτως. Το θέμα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφωνεί με, το, με τη σύμβαση και στην αιτιολόγησή του ο εισηγητής έδωσε πολύ συγκεκριμένους λόγους γιατί θα πρέπει να επικυρωθεί ένα τέτοιο πρωτόκολλο από τα κράτη-μέλη. Συνδέεται αυτό με τις πολιτικές απασχόλησης και την κοινωνική πολιτική και ο αγώνας αυτός εντός και εκτός της Ευρώπης απαιτεί αλληλεγγύη. Χρειαζόμαστε σαφείς κανόνες, χρειαζόμαστε διεθνή πρότυπα, τα οποία θα πρέπει να επικυρωθούν και να εφαρμοστούν και χρειαζόμαστε κοινή κατανόηση, διότι ο αγώνας ενάντια στην μαύρη εργασία μπορεί να πραγματοποιηθεί Μόνο από μια ενωμένη Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια τελική παρατήρηση της δικής μας πολιτικής ομάδας είναι ότι θα θέλαμε στα πρακτικά της σημερινής συνεδρίασης να καθίσατε σαφές ότι θεωρούμε απαράδεκτο ότι τα κράτη-μέλη ήδη ξεκίνησαν τις διαπραγματεύσεις για το πρωτόκολλο χωρίς προηγούμενη νομιμοποίηση από την Κομισιόν. Βρίσκουμε αμφισβητήσιμη την πρακτική αυτή και όπως και η Κομισιόν πιστεύουμε ότι κάτι τέτοιο μπορεί μόνο να αποτελεί εξαίρεση. Ζήταμε λοιπόν από το Προεδρείο της Επιτροπής μας να εκφράσει την αμφισβήτηση της διαδικασίας σε επιστολή προς το Συμβούλιο. Είμαι βέβαιη ότι το σύνολο της Επιτροπής Απασχόλησης συμφωνεί με τη θέση αυτή, διότι ε, εάν κάθε θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, κάνει ό,τι θέλει, ακόμα και σε τέτοιες περιπτώσεις ε, που επήγουν και που είναι προς όφελος όλων, τότε ε, παραβιάζουμε τους ε, κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα τέλος να ευχαριστήσω τον εισηγητή για μια πολύ καλή έκθεση και προσλέπουμε στην ε, συνέχιση της καλής συνεργασίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Χάρκινς και όδης από, από την Άλντε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όπως είπε και ο εισηγητής επικαιροποιούμε την τέταρτη σύμβαση και εδώ μιλούμε για την εφαρμογή της. Και στο πλαίσιο αυτό ζητούμε από τα κράτη-μέλη να αναπτύξουν μια εθνική πολιτική, ένα σχέδιο δράσεως, ώστε να εξασφαλίσουν την εξάλληψη της αναγκαστικής εργασίας και ελπίζουμε να έχουμε και άλλους φορείς και οργανισμούς ως συμβούλους. Χρειαζόμαστε μια εκστρατεία ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης ιδιαίτερα για τα θύματα, αλλά χρειαζόμαστε και ελέγχους πιο αυστηρούς και αποτελεσματικούς. Αυτό που είναι σημαντικό για τον πρωτόκολλο εδώ αυτό, για τα θύματα, πρέπει να αναλάβουμε ισχυρά μέτρα για την υποστήριξή τους και πρέπει να έχουν την δυνατότητα αποζημίωσης. Χρειαζόμαστε λοιπόν πρόσβαση, αποτελεσματική πρόσβαση σε ένα σύστημα αποζημίωσης και αντιστάθμισης ιδιαίτερα σε σχέση με τους μετανάστες ε, απασχολουμένους και ιδιαίτερα τις γυναίκες που είναι οι πιο εκτεθειμένοι και σε σχέση με τα όσα συμβαίνουν στην Νότια Μεσόγειο αυτή τη στιγμή πρέπει να το δούμε την κατάσταση αυτή διότι ένα από τα σχόλια που γίνονται είναι ότι πολύ συχνά τα έγγραφα δεν είναι τακτοποιημένα και μιλούμε για ανθρώπους που είναι απολύτως εκτεθειμένοι σε αυτή την κατάσταση πολλοί από αυτούς βρίσκονται σε ένα κενό αυτή τη στιγμή. και μπορούν να περιέλθουν σε μια τέτοια κατάσταση. Επίσης, δεν είναι μόνο εντός των δικών μας συνόρων που θα πρέπει να εξασφαλίζουμε ότι θα εφαρμόζεται αυτή η σύμβαση και θα την προσέχουμε, αλλά και εκτός των σύνορων μας. Και θα έλεγα, αναφερθήκαμε νωρίτερα και στο Κατάρ σε κάποιες άλλες περιπτώσεις, και ήδη είχαμε 1963 εργαζομένους που έχουν χάσει τη ζωή τους ή στην εργασία και έχουμε τις προϋποθέσεις για την καταναγκαστική εργασία όπως την ορίζει ο ΑΕΛΟ και επομένως σε σχέση με χώρες που δεν εφαρμόζουν τη σύμβαση αυτή θα πρέπει να το λάβει υπόψη της θεωρώ η Ευρωπαϊκή αυτό. Jim Lambert παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ τον εισηγητή για μια πολύ σαφή και πλήρη παρουσίαση σχετικά με το πρωτόκολλο αυτό του ΔΟΕ. Και σε σχέση με την ταχύτητα της πρόοδου, της στρατηγικής, συμφωνώ με τους προηγούμενους ότι αυτός θα πρέπει να είναι ο στόχος και όχι η προσθήκη άλλων στοιχείων ή σημείων που θα επιβράδυναν τη διαδικασία. Συμφωνώ επίσης ε, σχετικά με τις ομάδες αυτές πληθυσμού που είναι απολύτως ε, εκτεθειμένες ε, και όχι μόνο όπως αναφέρθηκε η συνάδελφος σε μετανάστες πολίτες τρίτων χωρών αλλά και Ευρωπαίους πολίτες δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως και τους άστεγους που πολύ συχνά έχουμε κρούσματα, περιπτώσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, και τη Σουηδία που χρησιμοποιούνται άστεγοι για να διοχετευθούν σε τέτοιου είδου ε, συστήματα. Χρειαζόμαστε λοιπόν πράγματι, μάλιστα υπάρχει και μια πρόσφατη μελέτη από το Βασίλειο, Τάφτ ε, σχετικά με πολύ ενδιαφέροντα πορίσματα. Πάντως θα συμφωνούσα απολύτως ε, με την προσέγγιση του εισηγητή, εμείς δεν πρόκειται να υποβάλουμε τροπολογίες. Ευχαριστούμε κυρία Αγκαία. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όπως και οι άλλοι συνάδελφοι. Συμφωνούμε και εμείς με την προσέγγιση του εισηγητή. Δεν πρόκειται να υποβάλουμε τροπολογίες ε, για το report και συμφωνούμε και με τις ε, προτάσεις που έγιναν ε, με, την όλη, με τον όλο προσανατολισμό. Απλώς μία-δύο παρατηρήσεις θα ήθελα να κάνω αν ε, θα μπορούσαν να είναι χρήσιμες. Ξεκινώντας από τη σύμβαση από το 1930, καταναγκαστική εργασία ορίζεται ως υπηρεσία που παρέχεται από άνθρωπο υπό απειλή, άνθρωπο που είναι περιορισμένη η ελευθερία του, και επομένως η υπηρεσία αυτή δεν παρέχεται οικειοθελώς. Πρόκειται για μια σαφέστατη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αυτό είναι κάτι που θα έπρεπε να υπογραμμίζουμε και να τονίζουμε. Αυτό δεν αφορά μόνο δυστυχώς στο παρελθόν αλλά και στο παρόν. 12 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο με τζίρο 32 δις δολάρια από αυτά από αυτήν την καταναγκαστική εργασία. Και θα ήθελα δύο προβλήματα να υπογραμμίσω. Καταρχάς το άρθρο 2 του πρωτοκόλου. Μεταξύ των μέτρων προλήψεως υπογραμμίζει την αναγκαιότητα να ε, υπάρξει ως ελέγχ... ελέγχων εργασιακών γιατί μόνο μέσω των ελέγχων θα μπορέσουμε να, καταγράψουμε και να επιλύσουμε το πρόβλημα και θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας και τις χώρες εκείνες στις οποίες κυρίως εμφανίζονται τα κρούσματα και τα προβλήματα αυτά διότι πλήγονται από την κρίση και επομένως έχουμε περισσότερες κατηγορίες του πληθυσμού πιο ευάλωτος σε τέτοια περιστατικά και κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να λάβει μέτρα για να προσθέσει τα να περιορίζει τα φαινόμενα, να αποκαθιστά τα θύματα, όπως και να παρέχει βοήθεια και στήριξη υπό άλλες μορφές. Στα πλαίσια των διεθνών ε, συνθήκων συμβάσεων και πρωτοκόλων, ε, αυτά τα αναγκαία ή κατάλληλα μέτρα είναι όρος που παραμένει ασαφής. Διότι κατά την άποψή μου αφήνουμε υπερβολική ελευθερία δράσεων και λιγμών και ο καθένας ε, ερμηνεύει και πράττει κατά το δοκούν. Μάλιστα ε, θα έλεγα μέχρι το σημείο να μην εφαρμόζονται καθόλου όλες αυτές οι συστάσεις. Ίσως λοιπόν και αυτές οι πτυχές θα έπρεπε να ελευθερθούν υπόψη. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ. Η κυρία Λιάσο Βιλιέκα. Ευχαριστώ πρόεδρε. η Είναι πολύ σημαντικό το πρωτόκολλο αυτό και υπάρχει μεγάλη ανάγκη να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των εργαζομένων και των μεταναστών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και για τους ίδιους τους πολίτες της Ένωσης. Θα πρέπει να γίνουν σεβαστά λοιπόν και τα θεμελιώδη δικαιώματα και να καταργηθεί το τράφικινγκ έχει μεγάλη σημασία το Κοινοβούλιο να υποστηρίξει την επικύρωση του πρωτοκόλου. Δεν θα συμφωνήσω όμως με την αιτιολόγηση του εισηγητή. Αναφέρεται στη Σύμβαση για Καταναγκαστική Εργασία μέσω εκμετάλλευσης, μέσω τράφικινγκ και συνδυάζει το θέμα αυτό με την απόσπαση των εργαζομένων. Αυτό δεν μπορούμε να το δεχτούμε εμείς. Αυτό είναι κάτι το οποίο γίνεται με νόμιμο τρόπο. Άλλωστε έχουμε υιοθετήσει μέτρα ε, τον προηγούμενο χρόνο για να σταματήσει η παραβίαση των νομικών ρυθμίσεων. Ήδη από το 2006 άλλαξε η βασική οδηγία και από τότε ισχύει το ότι η υποχρεωτική αμοιβή είναι ο υψηλότερος από τους μισθούς που θεωρείται ο κατώτατος σε κάθε χώρα. Δεν μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι 40.000 εργαζόμενοι που χρησιμοποιούν αυτό τον τρόπο εργασίας που είναι ιδιαίτερα ευνοϊκός θα θεωρηθεί ότι είναι στην κατηγορία του human trafficking και της εκμετάλλευσης. Δεν συμφωνώ με την αιτιολόγηση λοιπόν του κυρίου Λεϊαρίκ. Σας ευχαριστώ. Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής έχει το λόγο. Ο κύριος Διαλό από τη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης. Ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την έκθεσή του και για τη στήριξη στην πρόταση που συζητάμε. Να ευχαριστήσω λοιπόν και όλους τους εισηγητές. Τον Ιούνιο του 2014 η συνέλευση του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας και η τριμερής μεγάλη συνάντηση υιοθέτησε το νέο πρωτόκολλο στη Σύμβαση για την Καταναγκαστική Εργασία. Αυτό ήταν καρπός και της συμμετοχής των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε κάνει μεγάλες προσπάθειες για την υιοθέτηση του συγκεκριμένου μέσου. Μετά από την υιοθέτηση του μέσου αναλάβαμε δράση για την επικύρωση της πρότασης. Η πρόταση έγινε δεκτή τον μήνα Ιούνιο και η πρόταση για την απόφαση ε, του Συμβουλίου ήρθε το Σεπτέμβριο του 2014 όπως υπογραμμίζεται και στις διάφορες παρεμβάσεις που έγιναν, η καταπολέμηση της καταναγκαστικής εργασίας είναι σημαντική για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για εσωτερικούς και για εξωτερικούς λόγους. Είμαστε υπέρ της πρόθεσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των ανεκτών συνθήκων εργασίας και εσωτερικά και σε επίπεδο εξωτερικών σχέσεων. Το πρωτόκολλο θα συνεισφέρει σε μια καλύτερη προστασία των εργαζομένων στα διάφορα κράτη-μέλη της Ένωσης. Οι χώρες που θα επικυρώσουν το πρωτόκολλο αυτό συμφωνούν για την αποτροπή της χρήσης της καταναγκαστικής εργασίας και στα πλαίσια του τράφικινγκ, την βελτίωση της προστασίας των θυμάτων και την διευκόλυνση έβρεσης τρόπων αποκατάστασης. Λοιπόν, εμείς περιμένουμε με θετικό πνεύμα την σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έτσι ώστε να επικυρωθεί παγκόσμια και να εφαρμοστεί η σύμβαση αυτή. Αυτή η γρήγορη επικύρωση θα συνεισφέρει στην πρόληψη και των σημερινών μορφών αναγκαστικής εργασίας, παροχή προστασίας διεθνούς στα θύματα και ανάπτυξη της διεθνούς συνεργασίας. Ευχαριστώ. Thank you. Uh, the... Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Λεργιαρίκ. Euh, Ευχαριστώ πρόεδρε. Να ευχαριστήσω όλους όσους πήραν το λόγο. Διαπιστώνω με μία εξαίρεση μια ευρυτά τη συνένεση. Ε, ένας από τους συναδέλφους ε, αναφέρθηκε στο νόημα των λέξεων και στην αδυναμία των λέξεων όταν μεταφράζονται σε επίπεδο αρχών δικαίου. Συμφωνώ μαζί της. Όμως το κείμενο ως έχει θα αποτελούσε ένα θετικό βήμα για όσους είναι θύματα σήμερα της καταναγκαστικής εργασίας ή της υποχρεωτικής εργασίας. Νομίζω ότι αν εμείς υιοθετήσουμε την πρόταση αυτή, αν τα όργανα υιοθετήσουν την πρόταση αυτή, αυτό θα δώσει μια πιο ανθρώπινη ψυχή στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και ο, πόσο το έχει ανάγκη αυτό σήμερα. Λοιπόν, δεν θα απαντήσω νομίζω στην παρατήρηση την οποία έκανε εξ ονόματος σοσιαλιστικής ομάδας η συνάδελφος, εσείς θα το εκτιμήσετε αυτό. Κατανοώ αυτό το οποίο λέγει βέβαια. Δεν θα ήθελα όμως η κριτική αυτή, η παρατήρηση η δικαιολογημένη την οποία έκανε να μην δημιουργήσει νομολογία στη δουλειά μας. Συνεπώς εννοώ με αυτό ότι θα την υποστηρίξω. Αλλά αυτό εξαρτάται από εσά. Διευκρινίζοντας ότι σήμερα αυτό το οποίο έχει σημασία είναι να μπορέσουμε να στηρίξουμε και να υιοθετήσουμε το συγκεκριμένο κείμενο. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Η προθεσμία για τις τροπολογίες είναι η 18 Ιουνίου. 15 ή 16 θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή Απασχόλησης και έχει προγραμματιστεί το θέμα για την Ολομέλεια του Σεπτεμβρίου μετά τις θερινές διακοπές. Σας ευχαριστώ όλους για τη συνεισφορά σας. Προχωράμε τώρα στο σημείο 12 της ημερήσιας διάταξης. Μείωση των ανισοτήτων με ειδική εστίαση στην παιδική φτώχεια. Ελπίζουμε να είναι όλοι παρόντες. ώστε να μπορέσουμε να ακολουθήσουμε το πρόγραμμά μας. Θέλουμε λοιπόν να εξετάσουμε 309 τροπολογίες ε, που υποβλήθηκαν για το σχέδιο έκθεσης. Θα δώσω πρώτα το λόγο στην εισηγήτρια. Κυρία Τσούμπερ, παρακαλώ έχετε το λόγο. Obrigada, Sra. Presidente. Ε, Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου για την δουλειά που κάναμε μαζί με τους εσκιώδεις εισηγητές και τους προβουλευτές που υπέβαλαν τροπολογίες. Λάβαμε 309 τροπολογίες ε, για το θέμα της ε, παιδικής φτώχειας και νομίζω ότι αυτό αντικατοπτρίζει τη σημασία που δίνει η Επιτροπή μας στο θέμα αυτό. Μόλις την Πέμπτη ήταν, διατεθειμένες οι ήταν διαθέσιμες τροπολογίες σε όλες τις γλώσσες. Απομένει λοιπόν να γίνει κάποια δουλειά όσον αφορά την ανάλυση τους και τον συνδυασμό τους. Θα ήθελα ωστόσο να μοιραστώ μαζί σας κάποιες ιδέες. Καταρχάς, κάποια από τα σχόλια που λάβαμε ήταν θετικά και στηρίζουν πολλές από τις ιδέες μου και αποτελούν σημαντική συμβολή δεδομένου του ότι δεν έχουμε πάντα πολύ χώρο για την ε, έκθεση. Αρκετές από τις παρατηρήσεις που ακούσαμε λοιπόν ε, στόχο έχουν να εμπλωτίσουν το περιεχόμενο της έκθεσης. και ιδιαίτερα πιστεύω οι τροπολογίες που έχουν να κάνουν με τη βελτίωση της ποιότητας της στέγασης και έχουμε επίσης τροπολογίες για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας. Οι επισφαλείς θέσεις εργασίας για τους γονείς και η ανεργία έχουν ε, ε, ε, ήδη αναφερθεί στην έκθεση, αλλά ε, δεν έχουμε αναφερθεί στο θέμα της καταπολέμησης της αδήλωτης εργασίας. Αναφερόμαστε επίσης ε, στην βελτίωση των κοινωνικών υπηρεσιών των κρατών μελών. Κάποιες τροπολογίες προτείνουν ένα ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και μπορούμε να συμφωνήσουμε με αυτές. Άλλες τροπολογίες προτείνουν πρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα ιδιαίτερα βραχυπρόθεσμα μέτρα για τα κράτη-μέλη που βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Επίσης έχουμε τροπολογίες σχετικά με τον υπολογισμό του σχετικού επίπεδου φτώχειας Η έννοια αυτή έχει να κάνει με το ότι οι απόλυτε τιμέ δεν αντικατοπτρίζουν πάντα τι πραγματικέ ανάγκε. Είμαι λοιπόν ικανοποιημένη με τη σχετική τροπολογία. Έχουμε άλλες τροπολογίες που επιρρύπτουν την ευθύνη όχι μόνο στην κρίση, αλλά σε αυτούς που χρησιμοποιούν την κρίση ως δικαιολογία. Ελπίζω να μπορέσουμε να βρούμε ε, συμβιβασμό όσον αφορά την τροπολογία αυτή. Συχνά, μέτρα που έχουν εφαρμόσει κράτη-μέλη κατά τη διάρκεια της κρίσης οφείλονται στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Κατόπιν έχουμε κάποια θέματα πιο προβληματικά. η πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες, το δικαίωμα στην εκπαίδευση, θα πρέπει να παρέχεται δωρεάν σε όλους. Αυτή είναι μία από τις αρχές που έχουν εκφραστεί σε πολλαπλές τροπολογίες. Αυτό συνδέεται και με εκθέσεις της UNICEF. Τα παιδιά θα πρέπει να έχουν καθολική πρόσβαση στα δικαιώματά τους, στην εκπαίδευση και ε, στις υπηρεσίες υγείας, ασχετά από το εισόδημα των γονέων. Έχουμε περιθωριοποιημένες οικογένειες, οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνουν συγκεκριμένο είδος ε, κοινωνικής βοήθειας. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε τη, τα θεμελιώδη δικαιώματα για όλα τα παιδιά. Και τα παιδιά αυτά θα πρέπει να τα εξετάσουμε όχι μόνο στο πλαίσιο της οικογένειάς τους, θα πρέπει να εξετάσουμε και τις ε, ειδικέ τους ανάγκες. Κατόπιν έχουμε τις συστάσεις αναχώρα. Στο πλαίσιο της ε, ετήσιας έκθεσης ε, ανάπτυξης της Κομισιόν, της ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξωμήνου. Η πολιτική μας ομάδα δεν θα μπορέσει να στηρίξει τη σχετική τροπολογία, ίσως όμως να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμβιβασμό όσον αφορά κάποιες από τις σχετικές τροπολογίες. Υπάρχουν διάφορες τροπολογίες που θέλουν να διαγράψουμε την ιδέα ότι τα μέτρα λιτότητας αύξησαν τη βία, την οικογενειακή βία. συμπεριλαμβανομένης της βίας εις βάρος των παιδιών. Θα πρέπει να επικεντρωθούμε περισσότερο στο θέμα αυτό. Το έχουμε συμπεριλάβει, διότι βρήκαμε σχετικά στοιχεία σε μια σειρά εκθέσεων. Η αστάθεια εντός των οικογενειών ως αποτέλεσμα οικονομικών παραγόντων αποτελούσε έναν από τους βασικούς παράγοντες για την αύξηση της βίας. Αυτό με καλό τρόπο δεν δικαιολογεί τη, τη βίαιη συμπεριφορά. Είναι όμως επίμαχο το θέμα και θα πρέπει να το εξετάσουμε περαιτέρω. Άλλο θέμα στο οποίο δεν συμφωνούμε είναι οι τροπολογίες που προσπαθούν να μεταφέρουν το μήνυμα ότι Ε, τα κοινωνικά επιδόματα χρησιμοποιούν ε, από οικογένειες για άλλους λόγους από αυτούς ε, για τους οποίους δημιουργήθηκαν. Το ελάχιστο εισόδημα και τα κοινωνικά επιδόματα συχνά είναι ο μόνος τρόπος να επιβιώσει μια οικογένεια. Ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα είναι ότι τα εισοδήματα είναι τόσο χαμηλά ώστε να μην μπορούν να βγουν οι οικογένειες από, την κατάστασή τους και έτσι περιθωριοποιούνται. Υπάρχουν επίση τροπολογίε που υπονοούν ότι ο κόσμος δεν πληρώνει τον νίκη επειδή δεν θέλει, όχι επειδή δεν μπορεί, αλλά και αυτό δεν αντικατοπτρίζει τις ε, περιπτώσεις τις οποίες γνωρίζουμε εμείς. Κατόπιν υπάρχουν τροπολογίε. που θέλουν διαγραφή κάποιων σημείων ε, στην έκθεση. Η UNICEF και άλλες οργανώσεις στις εκθέσεις τους συμφωνούν ότι τα κοινωνικά επιδόματα δεν αρκούν για να μπορέσουν να ξεφύγουν οι οικογένειες αυτές από την φτώχεια. Τούτων λεχθέντων θα πρέπει να βρούμε συμβαστικές προτάσεις. Εργαζόμαστε προς τον στόχο αυτόν. Δεν έχουμε ακόμα τελική επιβεβαίωση. Σχεδιάζουμε όμως στις 30 Ιουνίου συνάντηση με τους σκιώδεις εισηγητές. Δεν ξέρω αν αυτή θα είναι η μόνη ε, συνάντηση που θα μας χρειαστεί, διότι έχουμε πολλές τροπολογίες. Θα ήθελα όμως και πάλι να ευχαριστήσω όλους για τη συνεισφορά τους και να επαναλάβω ότι είμαι στη διάθεσή σας ε, και προσβλέπω στη συνεργασία μαζί σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Σόιντροβα από το ΕΡΙΚΣ και όδηση παρακαλώ. Oui, merci. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χαίρομαι για τις πολλές συνεισφορές των συναδέλφων σε αυτήν την πολύ σημαντική γνωμοδότηση και σε σχέση με την θέση του ΕΛΚ να πω το εξή. Τα πιο σημαντικά ζητήματα προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση των φτωχών παιδιών είναι τα θέματα της οικογένειας, τα θέματα της ποιότητας της εκπαίδευσης. Στις τροπολογίες λοιπόν που υποβάλαμε, εκ μέρους του ΕΛΚ, αλλά και εκ μέρους των υπόλοιπων συναδέλφων της ομάδας, έχουμε επικεντρωθεί στα θέματα της οικογένειας, της ένδυας των παιδιών, που στην ουσία είναι το ίδιο θέμα με την ένδυα των οικογενειών τους, και επομένως πρέπει να εστιαστούμε στις ενισχύσεις προς τις βοήθειες μέσω επιδομάτων, μέσω κοινωνικών καταβολών, μέσω δραστικών μέτρων υπέρ των γονέων και νομίζω αυτή είναι η διαφοροποίηση που θα έβρισκα μεταξύ των τροπολογιών που προτείναμε και της ε, τοποθέτησης ε, του εισηγητή. Και δεν θα συμφωνούσα σχετικά με τις δημοσιονομικές ευθύνες ε, για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων και της φτώχεια μεταξύ των παιδιών. Νομίζω ότι πρόκειται για μια τοποθέτηση υπερβολικά ιδεολογική. Πρέπει να υπογραμμίζουμε την ευάλωτη κατάσταση των παιδιών που προέρχονται από περιθωριοποιημένες κοινωνικές ομάδες όπως ε, το υπογράμμισε και η συνάδελφος Γιωτινιάνσκα. Ε, Επίσης θα ήθελα να υπογραμμίσω το θέμα της αυξανόμενης τάσης της εγκατάλειψης ε, των σχολείων και το οποίο έχει σχέση και με τις δυσμενείς προοπτικές ε, των παιδιών. Των παιδιών δηλαδή που απειλούνται από το φάσμα της φτώχειας. Αυτές είναι οι δικές μας προτάσεις. Ε, περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον την συζήτηση αυτή και είμαι βέβαιο ότι θα μπορέσουμε να εξεύρωμε συμβιβαστικές θέσεις ώστε να έχουμε μια πιο κοινή θέση πιο συμπεφωνημένη διότι πιστεύω ότι η γνωμοδότηση αυτή, η έκθεση αυτή θα μπορούσε να είναι η φωνή και το μήνυμα του Κοινοβουλίου προκειμένου να αλλάξει η κατάσταση. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Λεκινησιούτε, ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την παρουσίαση των τροπολογιών και εμείς είχαμε υποβάλει από πλευράς της ομάδας μας για νέα μέτρα που ενδεχομένως θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν στην καταπολέμηση των φαινομένων αυτών. Εμείς είχα, είχαμε προτείνει μάλιστα και ένα ταμείο εγγύησης για τα παιδιά αυτά ακριβώς ώστε να μπορεί να έχει πρόσβαση το καθένα από αυτά τα παιδιά στις στοιχειώδεις και απαραίτητες υπηρεσίες ε, υγείας βασικής κοινωνικής καλύψεως που θα ήταν αντίστοιχο μέσω με εκείνο της πρωτοβουλίας για τους νέους. Εμείς θεωρούμε ότι τα κράτη-μέλη θα έπρεπε να αναπτύξουν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο καταπολέμησης της στόχιας των ε, παιδιών με εγγυήσει και δίνοντας τη δυνατότητα στους γονείς των παιδιών αυτών να βγουν από την περιθωριοποίηση και να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Επίσης καλούμε τα κράτη-μέλη να αναλάβουν να προχωρήσουν και στις κατάλληλες επενδύσεις εφαρμόζοντας και τις ε, συστάσεις της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία και εκείνη θα πρέπει να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της προκειμένου τα κρατημέλη να επιτηρούν ετησίως και να υποβάλουν τακτικές εκθέσεις σχετικά με την πρόοδό του στα κρατη Θεωρούμε ότι ε, επίσης ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τα διαρθρωτικά ταμεία της Ερωικής Ένωσης ώστε όλα αυτά τα παιδιά να μπορούν να έχουν ένα αποδεκτό επίπεδο ποιότητας ζωής και να έχουν πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες και μάλιστα σε ποιοτικές υπηρεσίες ώστε να ξεφύγουν από την παγίδα αυτή της φτώχειας. Θεωρούμε επίσης ότι η Κομισιόν θα πρέπει να έχει και ένα συμπληρωματικό στόχο στα πλαίσια του Ευρώπη 2020, δηλαδή την μείωση της ε, φτώχειας μεταξύ των παιδιών και του κοινωνικού τους αποκλεισμού. Θα πρέπει, θεωρούμε, να ευαισθητοποιηθούν όλα τα κρατη επί του προβλήματος αυτού και καλούμε την Κομισιόν όταν συντάσσει τις προόδους των κρατών μελών της δημοσιονομικές να εγγράφει και ένα συγκεκριμένο στόχο, αυτόν εδώ. Θα πρέπει στα παιδιά αυτά να προσφέρονται και συγκεκριμένα προγράμματα δραστηριότητα στα πλαίσια της παιδείας ώστε να εγγυόμαστε, ώστε να μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι όλα τα παιδιά θα έχουν πρόσβαση στο απαραίτητο σχολικό υλικό, αλλά και στις μεταφορές από και προς το σχολείο. Εμείς θεωρούμε ότι η Κομισιόν θα πρέπει να έχει μια στρατηγική καταπολέμηση στη στόχια των παιδιών. Η οποία να εστιάζεται κυρίως στη ρίζα του φαινομένου αυτού, στην προέλευση του. Θα πρέπει λοιπόν να εξασφαλίζει, να διασφαλίζει μάλλον κάποιες κατώτατες κοινωνικές ε, εγγυήσει και ένα κατώτατο εισόδημα για τις οικογένειες των παιδιών αυτών γιατί μιλούμε για φαινόμενα τα οποία είναι αποτέλεσμα αυτής της παρατεταμένης κρίσεως και των μέτρων λιτότητας και αυξάνεται συνεχώς όχι μόνο η φτώχεια των οικογενειών αλλά και των παιδιών ως απόρρια όλων αυτών των πολιτικών. Πρέπει λοιπόν να κινητοποιηθούν τα απαραίτητα κοινωνικά μέσα, επιδόματα και κονδύλια προκειμένου να ε, ενισχυθούν, να υποστηριχθούν αυτές οι ομάδες πληθυσμού και ιδιαίτερα τα παιδιά. Δεν, δεν θεωρώ ότι πρέπει να αναλωνόμαστε εδώ μεταξύ κομματικής φύσεως υποθετήσεων, θα πρέπει όλοι να συνεργαστούμε και να βρούμε συνενετικές απόψεις και συμβαστικές λύσεις ώστε να επιτύχουμε αποτελέσματα στο πεδίο, απτά αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν βλέπω εδώ τον σκιώδη των συντηρητικών. Αυτό σημαίνει ότι θα περάσουμε απευθείας στον πρόσωπο τον σκιώδη συγγητή της Άλντε την σκιώδη συγγήτρια της Άλτα. Κυρία Τόμ, το θέμα αυτό είναι πολύ ευαίσθητο και σημαντικό. Βλέπουμε ότι ιδιαίτερα στα νεότερα κράτη-μέλη υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα παιδικής εργασίας. Στην Εστονία πάνω από το 10% των παιδιών ζουν κάτω από συνθήκες φτώχειας. Εμείς ζητήσαμε από το Κοινοβούλιο να καταθέσει ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την καταπολέμηση της φτώχειας που χτυπάει τα παιδιά. Αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας είναι η εφαρμογή και για τα παιδιά των ελαχίστων κοινωνικών κανόνων. Εξ ονόματος λοιπόν της ομάδας των φιλελευθέρων καταθέσαμε κάποιες ε, τροπολογίες στην έκθεση δεν θα αναφερθώ σε όλες αυτές. Για τους έφραυτους πληθυσμούς, όπως παιδιά μετανοστών, γυναίκες, Ρωμά και ανθρώπους οι οποίοι ανήκουν σε συγκεκριμένες μειονότητες και υφίστανται τον κοινωνικό αποκλεισμό περισσότερο. Ελπίζω να συνεχίσουμε λοιπόν με σωστό τρόπο να μην δώσουμε πολιτικής φύσης μάχες και ίσως, ίσως λέω να πετύχουμε. You, ε, Jean Green's Shadow. Η σκιώδη των πρασίνων Λάμπερτ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τον εισηγητή. Εμείς έχουμε συνεισφέρει τα μάλα στον μεγάλο αριθμό των ε, τροπολογιών που έχουν κατατεθεί, αλλά νομίζω ότι ακολουθούμε την ε, πορεία την οποία δείχνει η έκθεση. Υπάρχουν πολύ καλά υλικά μέσα σε αυτή την πρόταση. Προς το παρόν όμως υπάρχει δυνατότητα βελτίωσης. Το θέμα είναι λοιπόν πώς θα μπορέσουμε να εντάξουμε τις προτάσεις αυτές και στα πλαίσια του λεγόμενου εξαμήνου. Έχουμε κάποιες ανησυχίες τις οποίες προσπαθούμε να βάλουμε στην έκθεση. Ξέρετε εσείς ότι μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ το θέμα των κοινωνικών επιπτώσεων των μέτρων που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια της κρίσης έτσι ώστε να καταλάβουμε πώς τα μέτρα αυτά έχουν λειτουργήσει στα πλαίσια της στρατηγικής καταπολέμησης της φτώχειας και κατά πόσο έχουν αυξήσει τη φτώχεια. Λοιπόν, αυτού του είδους η αξιολόγηση για μας είναι ένα κομβικό μέσο το οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο πρέπει να χρησιμοποιήσει. Υπάρχει επίσης το θέμα των, της στρατηγικής ε, για τους αστέγους. Είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να μας απασχολήσουν. και στα πλαίσια της προσπάθειας καθιέρωσης του ελάχιστου κοινωνικού εισοδήματος ή και χρήσης όλων των δυνατών μέσων Υπάρχει το θέμα της συμμετοχής των ίδιων των παιδιών στις συζητήσεις για το μέλλον τους και ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών. Έχει μεγάλη σημασία όταν μιλάμε για τα δικαιώματα των πολιτών να διασφαλίσουμε και τη συμμετοχή τους στις συζητήσεις αυτές. Προσβλέπουμε λοιπόν στην συνάντηση των σκιωδών και ελπίζω να γίνουν μαγικά και να συρρυκνωθεί ο αριθμός των τροπολογιών. Νομίζω ότι εντάσσονται όλες σε ένα κοινωνικό πλαίσιο και αυτό είναι κάτι το οποίο έτσι κι αλλιώς μας απασχολεί ακριβώς το κοινωνικό πλαίσιο για το αν οι βοήθ, οι οικογένειες στηρίζονται στην προσπάθειες τις οποίες κάνουν. Ιδιαίτερα οι κατηγορίες αυτές που περιθωριοποιούνται και ζουν εκτός των συστημάτων έτσι όπως λειτουργούν σήμερα. Θα πρέπει και αυτή την κατηγορία των παιδιών να μας απασχολήσει. Ευχαριστώ πολύ. Αντζέα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ την κυρία Ζούμπερ για την προσπάθεια που έκανε και για τη διαθεσιμότητα που επέδειξε. Εμείς στρέψαμε την προσοχή μας στην, ε, στις που δημιουργούν αυτό το πρόβλημα στην παιδική ηλικία. Είναι, υπάρχει ανάγκη να δράσουμε πλέον, όχι τόσο στα, σε σχέση με τις συνέπειες, αλλά σε σχέση με τις αιτίε. Η παιδική φτώχεια είναι καρπός της μακράς ανεργίας, την οποία βιώνουν οι διάφορες οικογένειες. Είναι επίσης πολλές φορές καρπός της οικονομικής κρίσης, η οποία εδώ και αρκετά χρόνια χτυπά πολλά, πολλές περιοχές της Ευρώπης και οδηγεί σε σοβαρότατες συνέπειες οι οποίες ε, χαρακτηρίζουν τις οικογένειες, χτυπούν τις οικογένειες, ιδιαίτερα τις πιο ευάλωτες και τα χειρότερα επιφυλάσσονται για τα παιδιά. Ακούγεται παράλογο, αλλά υπάρχουν ε, σοβαρές μελέτες οι οποίες λέγουν ότι μία από τις ασθένειες τις οποίες βιώνουν τα παιδιά και είναι η ραχίτιδα την οποία παθαίνουν λόγω της κακής διατροφής. Είναι απαράδεκτο τον 21ο αιώνα στην Ευρώπη να υπάρχει έστω και ένα παιδί που να είναι ραχιτικό επειδή δεν τρώει σωστά. Λοιπόν, πρέπει να σταματήσουμε τα λόγια και να βοηθήσουμε όλες αυτές τις εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά που δεν έχουν σωστή διατροφή. Απαιτείται λοιπόν άμεση δράση, ισχυρή δράση, χωρίς καμία πρόκληση, χωρίς κανένα δισταγμό, συγγνώμη, και νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας θα πρέπει έστω και μέσω του ελάχιστου εισοδήματος να βοηθήσουμε τα παιδιά αυτά. Δεν είναι υποβοηθητικά τα μέτρα αυτά, δεν είναι υποσπάθεια να τα καλύψει η πρόνοια, αλλά να μπορέσουμε να καταστήσουμε ικανούς τους γονείς να διατρέφουν σωστά τα παιδιά τους. Εμείς πολλές φορές αντιμετωπίζουμε όλα αυτά τα μέτρα με οικονομικό και νομισματικό τρόπο, αλλά εγώ όταν αναφέρομαι σε υποστήριξη σε οικογένειες που έχουν δυσκολίες, αναφέρομαι περισσότερο σε υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται με δωρεάν τρόπο. Σαν παράδειγμα να μην έχουν δίδακτρα, να πληρώνονται ε, τα έξοδα μεταφοράς. Υπάρχουν, εν πάση περιπτώσει, τρόποι που θα βοηθήσουν τις οικογένειες αυτές να δράσουν με σωστό τρόπο. Η εκπαίδευση είναι και αυτό κεφαλαιόδες σημείο του τρόπου δράσης μας. Είναι απαραίτητο να υπάρξει εγγυημένη δυνατότητα εκπαίδευσης και τα παιδιά τα οποία ζουν σε κατοστάσεις κινδύνου περιθωριοποιημένα να μην φεύγουν από το σχολικό κύκλωμα αλλά να υπάρχουν ειδικέ δράσεις που προστατεύουν, καθοδηγούν τα παιδιά αυτά και δεν τα αφήνουν να φύγουν από τη σχολική διάρκεια πρόωρα. Για αυτά τα παιδιά πρέπει λοιπόν να δράσουμε με στοχευμένο τρόπο, σε αυτά τα παιδιά πρέπει να στραφεί η προσοχή μας για μια εκπαίδευση δωρεάν, εγγυημένη, ποιοτική και οι κοινωνικές υπηρεσίες και στον τομέα της παιδείας και στον τομέα της υγείας για τις ε, κατηγορίες τις περιθωριοποιημένες που ζουν μέσα στη φτώχεια που είναι σε κίνδυνο για αυτές τις κατηγορίες θα πρέπει να ενισχυθούν τα μέτρα αυτά. Θα συμφωνήσω με την συνάδελφο του Σοσιαλδημοκρατικής Ομάδας. Πράγματι δημιουργήσαμε ένα ταμείο για τους νέους, για να μπορέσουμε να δώσουμε νέες δυνατότητες στους νέους να δουλέψουν Προσπαθήσαμε να οργανώσουμε κάτι σημαντικό επίσης και για τα παιδιά. Είναι ηθικό μας καθήκον. Το καθένας από εμά θα πρέπει να νιώσει αυτή την τεράστια ευθύνη έτσι ώστε να προστατεύσουμε και το τελευταίο από τα παιδιά της Υπήρου μας. Γιατί στην ουσία τα παιδιά είναι ο καθρέφτης της δουλειάς μας, είναι η εικόνα που δείχνει αν δουλεύουμε καλά ή αν δουλεύουμε άσχημα. Ευχαριστώ λοιπόν την συνάδελφο και είμαστε διατεθειμένοι να συνεργαστούμε μαζί της αν και σε ορισμένα θέματα δεν υπάρχει πια περιθώριο. Ή θα πρέπει να δράσουμε άμεσα ή θα πρέπει πράγματι να αναρωτηθούμε γιατί λειτουργούμε. Ευχαριστώ πρόεδρε, λέει η κυρία Ριμπέιρο. Πρόκειται ένα θέμα που πρέπει να μας απασχολήσει πολύ. 26 εκατομμύρια παιδιά φαίνεται ότι απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό και φτώχεια. Είναι υπερβολικά μεγάλο το μέγεθος για να είμαστε αδιάφοροι. Η Κομισιόν θα πρέπει να εξασφαλίσει την ευρύτερη δυνατή συνένεση και πραγματικά ε, θα έλεγα και προς την εισηγήτρια ότι πρέπει να βρούμε συνενέσεις εδώ. Και εδώ μιλούμε για επιπτώσεις και για τις μελλοντικές γενναίες. Η ασφάλεια και η υγεία των παιδιών αυτών θα πρέπει να εξασφαλιστεί και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αναλάβουν μέτρα προς τις πιο περιθωριοποιημένες ή ευάλωτες οικογένειες. οι οικογένειες θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας και τα παιδιά θα πρέπει να έχουν πρόσβαση ε, στην παιδεία και την κοινωνική υποστήριξη. Θα πρέπει οπωσδήποτε να στηρίζουμε τους νέους και τα παιδιά της Ευρωπαϊκή Ένωσης με μέσο μακροπρόθεσμους στόχους καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού. Θα πρέπει να αναπτύξουμε μια οικονομική πολιτική αν θέλετε για τις οικογένειες και για τους νέους και τα παιδιά. Υπάρχουν κοινωνικά προγράμματα, είναι αλήθεια, αλλά θα πρέπει να εφαρμόζονται καταλήλως, θα πρέπει να τα παρακολουθούμε και να τα ελέγχουμε, θα πρέπει να καταπολεμήσουμε όλα αυτά τα φαινόμενα περιθωριοποίησης και αποκλεισμού. Έχουν υποχρέωση τα κράτη-μέλη να αναπτύξουν συμφωνίες συνεργασίας με όλους εκείνους τους οργανισμούς και τους φορείς που είναι που προσπαθούν να υποστηρίξουν την κατάλληλη κοινωνική ένταξη αυτών των οικογενειών και αυτών των ομάδων. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλους τους δυνατούς πόρους. Κάνουμε έκκληση στα κράτη-μέλη και, και στην Κομισιόν να δημιουργηθούν διακρατικά δίκτυα καλύπτοντας και τις απόμακρες περιφέρειες. Θα πρέπει να καλύψουμε το σύνολο του πληθυσμού των παιδιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Η κυρία ε, Ζούμπερ θα ήθελε να, να κλείσει κάπως. Ναι, πολύ σύντομα πρόεδρε να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για τις συνεισφορές τους Θα έχουμε και τις επόμενες συναντήσεις με τους Κιώδης και θα το ξανασυζητήσουμε. Ε, έχω την εντύπωση ότι η πλειοψηφία των προτάσεων που υπευλήθησαν ακολουθούν τη γραμμή που υπερασπίζεται και η δική μας ομάδα. Νομίζω ότι έχουμε μια κοινή κατεύθυνση δηλαδή. Υπάρχει όμως κάτι στο οποίο θα ήθελα να αναφερθώ συγκεκριμένα Και εδώ δυσκολεύτηκα και εγώ προκειμένου να συντάξω το κείμενο σχετικά με τις αιτίες και τα αποτελέσματα. Εδώ λέμε πράγματα μάλλον παρατηρούμε πράγματα τα παρατηρούμε και τα καταγράφουμε και δεν τα επινοούμε σχετικά με τις αιτίες των φαινομένων αυτών. Εγώ προσπάθησα να βρω όλες τις ε, πληροφορίες που μπορούσα χωρίς να έχω κανενός είδους ιδεολογική αν θέλετε κατεύθυνση. Πρόκειται για δεδομένα και πληροφορίες που καταγράφουν το φαινόμενο της φτώχειας μεταξύ των παιδιών. Οι περικοπές των κοινωνικών υπηρεσιών, των επιδομάτων, η κατάσταση που βιώνουν οικογένειες οι οποίες έχουν ε, γονείς δηλαδή που έχουν απολυθεί δεν είναι πράγματα που έχω επινοήσει δεν είναι πράγματα που είναι φανταστικά αν κάνουμε μια διάγνωση των αιτιών που οδηγούν σε αυτά τα φαινόμενα πρέπει αναγκαστικά να αναφερθούμε σε αυτά τα πράγματα θεωρώ λοιπόν ότι ναι πρέπει να το συζητούμε ως φαινόμενο καθεαυτό αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να συζητούμε για τις αιτίες του φαινομένου. Το να περιοριζόμαστε σε μία διακήρυξη αρχών και αξιών επί της οποίας προφανώς όλοι εδώ συμφωνούμε δεν έχει νόημα. Εδώ χρειαζόμαστε να βρούμε τα αίτια και μετά να πούμε τι κοινωνικά μέτρα θέλουμε να εφαρμόσουμε προκειμένου να επιδιορθώσουμε τα αποτελέσματα και τα φαινόμενα αυτά. Πάντως θα το ξανασυζητήσουμε και στις συναντήσεις και με τους Χιώδης και τις υπόλοιπες. Σας ευχαριστώ λέει Πρόεδρος για μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για τη φτώχεια των παιδιών. Το, το κάναμε αυτό μια-δύο φορές τα τελευταία χρόνια και προσμένουμε, περιμένουμε με ενδιαφέρον τα αποτελέσματα αυτή ήταν και η κατεύθυνση των 309 τροπολογιών 15 και 16 Ιουλίου αναμένεται η υποβολή και πάμε στο 13 τώρα, νομίζω το τελευταίο στην διάταξη για την κοινωνική επιχειρηματικότητα και κοινωνική καινοτομία για την καταπολέμηση της ανεργίας. Είναι οι 180 τροπολογίες για την γνωμοδότηση πρωτοβουλίας της κυρίας Βερόνικα Λόπεθ Φοντανιέ στην οποία δίνω και λόγο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Πράγματι έχουμε 180 τροπολογίες αλλά πολλές από αυτές, να σας καθησυχάσω, πάνε προς την αυτή κατεύθυνση. Η δουλειά είναι αρκετά προχωρημένη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω λοιπόν πρώτα απ' όλα τους συναδέλφους και ιδιαίτερα τους Κιώδης για την ε, συνεργασία και το πνεύμα το επικοδομητικό με την, υπό το οποίο έγινε αυτή. Ήδη συζητήσαμε 20 τροπολογίες και συμφωνήσαμε που θα υποβληθούν στην επόμενη συνάντηση της Επιτροπής. Η δουλειά δεν είναι τόσο περίπλοκη θα μπορούσα να πω καθότι η πλειοψηφία που σας έλεγα των τροπολογιών πηγαίνουν στη βελτίωση της κοινωνικής οικονομίας, της αναγνώρισής της και της σημασίας της όχι μόνο υπό την κοινωνική αλλά και υπό την περιβαλλοντική έννοια ή την εδαφική. Αυτά σημαίνουν ότι η γνωμοδότηση βελτιώνεται ουσιαστικά. Πολλές από τις τροπολογίες προς την κατεύθυνση αυτήν πάνε ως και ως προς το σχετικό στίγμα για κάποιες εταιρείες και προσπαθούμε να προωθήσουμε σε όλα τα επίπεδα την πρόσβαση στη χρηματοδότηση και να έχουμε μια συμπεφωνημένη εικόνα για τις επιχειρήσεις αυτές οι οποίες θα πρέπει να καταστούν ελκυστικότερες για τους νέους. Πρέπει λοιπόν να προωθούμε την καινοτομία και την κοινωνική αν θέλετε εκπαίδευση καλύπτουμε την κοινωνική επιχειρηματικότητα και ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα είναι η απτή αναφορά στις θεματικές αυτές. Κάποιες από τις τροπολογίες προχωρούν πιο πέρα από τι κάνουμε εντό του κειμένου για τις ε, δημόσιες επενδύσεις, για τις δημόσιες δαπάνες που είναι ναι θετικά αν θέλετε σημεία αλλά τα οποία δύσκολα ενσωματώνονται στην ε, γνωμοδότηση και είναι η μόνη ομάδα τροπολογιών για τις οποίες θα ζητήσω ε, την ε, ψηφοφορία. Ένα άλλο σημείο όμως το οποίο βοηθά και συνεισφέρει είναι του κυρίου Μπέκερ για την αναγκαιότητα ε, δουλειάς επί των ρυθμιστικών κειμένων ε, που διέπουν την επιχειρηματικότητα αυτού του είδους. Έχω επίσης ε, για την ε, τροπολογία της 158 της κυρία Τζέα όπου ζητάει συγκεκριμένο δημοσιονομικό κονδύλιο ε, στα πλαίσια του κοινωνικού ταμείου. Όπως τα ξέρετε, αυτό δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε αυτή τη στιγμή παρότι θα μας ικανοποιούσε να μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε διότι αναφέρεται σε άλλες συμπεφωνημένες περιοχές. Το κοινωνικό λοιπόν ταμείο είναι, έχει κάποιους περιορισμούς στις δυνατότητες που έχουμε να το χρησιμοποιήσουμε αυτή τη στιγμή. Τώρα, εδώ έχουμε ευθείε συνέπειε της κρίσεως. 1,3 εκατομμύρια θέσεων απασχόληση μεταξύ του 2009 και 2013 έχουμε στον τομέα αυτών και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και γι' αυτό θεωρώ ότι η γνωμοδότηση αυτή θα πρέπει να επιτύχει την ευρύτερη δυνατή συνένεση και θα πρέπει να στηρίξουμε τις ε, επιχειρήσεις αυτές που σε αυτή τη στιγμή της κρίσεως ήταν αυτές που απεδείχθησαν οι πιο ανθεκτικές. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, Σας ευχαριστώ. Ήταν μια καλή εισαγωγή στη συζήτηση. Θα δώσω τώρα το λόγο στον εκπρόσωπο των Σοσιαλδημοκρατών. Ο Φέι. Ευχαριστώ την Λόπε Φοντανιέ. Είχαμε μια καλή πρώτη συνάντηση. Νομίζω ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία στις βασικές συμβιβαστικές προτάσεις που έκανε. Τώρα για τις διάφορες τροπολογίες να πω ότι μπορούμε να υποστηρίξουμε εμεί τη μεγάλη τους πλειοψηφία γιατί ορίζουν με σωστό τρόπο όλα τα θέματα που καλύπτονται από το αρχικό κείμενο. Εμείς θεωρούμε ότι οι επιχειρήσεις αυτές της κοινωνικής οικονομίας στηρίζουν την τοπική κοινωνία και διευκολύνουν την χρηματοδότησή τους με τον τρόπο αυτό και σε τοπικό επίπεδο και σε εθνικό επίπεδο. Εμείς θεωρούμε ότι η κοινωνική γενικά ε, επιχείρηση και η κοινωνική επιχειρηματικότητα πολλές φορές γεφυρώνει τα κενά που υπάρχουν σε σχέση με συγκεκριμένες κοινωνικές κατηγορίες. Υπογραμμίζουμε τον τρόπο με τον οποίο θέλουν να βελτιώσουν τις παροχές υπηρεσιών. Είναι κάτι που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη όταν συμμετέχουν σε διαδικασίες διαγωνισμών και προμηθειών του δημοσίου. Προσπαθούμε εμείς να διασφαλίσουμε το ύψιστο δυνατό επίπεδο νομικής αναγνώρισης υιοθετώντα τους ορισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια του προγράμματος EASY. Αυτό έχει συζητηθεί και στην τελευταία συνάντηση των συντονιστών. και τίθεται και το θέμα φυσικά της κοινωνικής επένδυσης, της έννοιας της κοινωνικής επένδυσης που διευκολύνει κατά πολύ α, τις συζητήσεις μας. Κλείνοντας θα πω ότι ελπίζω να στηρίξετε την 116 που καταδικάζει την έλλειψη ενδιαφέροντος που δείχνει η στρατηγική ψηφιακή της Επιτροπής στην κοινωνική οικονομία και τις επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονομίας. Αυτό είναι κάτι το αρνητικό. Γιατί τίποτα από ό,τι φαίνεται δεν μπορεί να βοηθήσει αυτούς οι οποίοι έχουν συγκεκριμένα προβλήματα αναπηρίας, σαν παράδειγμα, να καλύψουν τις κοινωνικές τους ανάγκες. Μιλάμε για εδώ μεγάλο έλλειψη οράματος από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας ευχαριστώ πολύ. ο σκιώδης των συντηρητικών. Θέλετε το λόγο. Θα ακούσουμε πρώτα την κυρία Χάρκιν από την Άλτε και κατόπιν θα επιστρέψουμε στο ECR. Ευχαριστώ. Θα είμαι πολύ σύντομη. 30 δευτερόλεπτα. Συγχωρήστε με. Ευχαριστώ πολύ. Είχαμε πολύ καλή συνάντηση των σκιωδών εισηγητών. Υπάρχει μια σειρά συμβιβασμών που θα πρέπει να αναδιατυπωθούν, αλλά γενικά υπήρχε συμφωνία για πολλές από τις ε, ιδέες που υποβλήθηκαν. Το καθεστώς παρεκκλήσεων ε, νομίζω ότι λύθηκε, άργησα να φτάσω. Συμφωνώ με τους σοσιαλιστές όσον αφορά την διατύπωση για το πρόγραμμα ε, Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να χρησιμοποιήσουμε την ιδέα αυτή στην έκθεση και ε, δαπανίσαμε αρκετό χρόνο στη διατύπωσή της. Κάποιες από τις ε, τροπολογίες της Άλγα είχε να κάνει με τις κοινωνικές ανισότητες, ε, το ξεκλείδωμα του δυναμικού όσον αφορά τις θέσεις απασχόλησης και το θέμα των δημοσίων συμβάσεων που δεν ξέρω αν είναι πρόβλημα σε άλλα κράτη-μέλη αλλά στη δική μου χώρα συχνά οι δημόσιες συμβάσεις είναι σχεδιασμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να αποκλείουν τις μικρότερες εταιρείες, όχι απαραίτητα λόγω του μεγέθους, αλλά λόγω των απαιτήσεων. είναι πιο εύκολο για τους υπεύθυνους ε, ότι πρέπει να ασχοληθούν μόνο με ε, έναν δύο. Ε, αλλά αυτό σημαίνει ότι αποκλείονται οι μικρότερες επιχειρήσεις ε, με την πρώτη ματιά. Και τέλος ε, να πω και πάλι ότι συμφωνώ ότι το πακέτο κοινωνικών ε, επενδύσεων θα πρέπει να προωθηθεί και η κοινωνική οικονομία να παίζει σημαντικότερο ρόλο στο συνολικό πακέτο κοινωνικών επενδύσεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Κρασντέσκη που είναι ισχυώδης ε, των συντηρητικών. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι είχαμε πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση πάνω στις τροπολογίες. Ιδιαίτερα πολύτιμες ε, είναι οι τροπολογίες, ε, οι συμβιβαστικές κάπα και μη που αναφέρονται στην ανάγκη για καλύτερη πληροφόρηση. Στην συμβιβαστική μη αναφερόμαστε στους παράγοντες της κοινωνικής οικονομίας και δεύτερον στην συμβιβαστική τροπολογία K λέμε ότι θα πρέπει να τονίσουμε την πολυμορφία στην κοινωνία και τις διαφορετικές ανάγκες των διαφόρων κοινωνιών. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη μας τα διαφορετικά πλαίσια. Επιπλέον, θα ήθελα να πω ότι στην συζήτησή μας υπήρχε η τάση να αντιπαραθέτουμε την κοινωνική οικονομία απέναντι στις παραδοσιακές επιχειρήσεις. Μιλάμε δηλαδή για επιχειρήσεις που δεν έχουν αποκλειστικό στόχο το κέρδος. Έχουν μια επιπλέον αποστολή. Πιστεύουμε ότι είναι σημαντική η προσθήκη αυτή, δεν θα πρέπει όμως να θεωρήσουμε ότι οι κοινωνικές επιχειρήσεις μπορούν να αντικαταστήσουν τις κανονικές επιχειρήσεις. Θα ήταν υπερβολικό δηλαδή να τις θεωρήσουμε πρότυπο για το σύνολο της οικονομίας. Είναι βέβαια πολύ σημαντικό το θέμα της κοινωνικής οικονομίας και συμφωνώ με αυτό. Ευχαριστώ κυρία Λαούρα Ατζέα, παρακαλώ. Ε, Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ και την εισηγήτρια. Έχει λάβει υπόψη τη τις προτάσεις τις οποίες έχουμε καταθέσει. Θεωρώ ότι η κοινωνική επιχειρηματικότητα είναι ένα ικανό μέσο το οποίο σε μια φάση κρίσης όπου μειώνεται η παραγωγή, όπου η ζήτηση και η προσφορά πράγματι ελαττώνονται, μπορούν να βοηθήσουν έτσι ώστε να ελαφρυνθούν τα αρνητικά αποτελέσματα της κρίσης ιδιαίτερα στον τομέα της απασχόλησης. Και αυτό όχι μόνο για να καταπολεμήσουμε την ανεργία των νέων, αλλά κυρίως για να καταπολεμήσουμε τη μακρόχρονη ανεργία. Και γι' αυτό εκτιμήσαμε δεόντως την προσοχή η οποία δόθηκε και στη δική μας τροπολογία. Ένας από τους βασικούς στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020 είναι η μείωση κατά 75% ε, στον τομέα της εργασίας, της απασχόλησης. Νομίζω ότι θα πρέπει να στοχεύσουμε ψηλότερα και να αναζητήσουμε νεότερους δρόμους, καινοτόμους δρόμους για να δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης. Είναι προφανές ότι τα παλαιά μέσα δεν είναι πλέον αποτελεσματικά. Υπάρχει επίσης μια άλλη διάσταση στην οποία πρέπει να σταθώ. Η ανάγκη που υπάρχει τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν μέτρα τα οποία να στηρίζουν αποτελεσματικά ε, ε, να δοθούν κίνητρα με λίγα λόγια στις κοινωνικές αυτές επιχειρήσεις. Γιατί αυτό δεν θίγει μόνο αυτούς οι οποίοι έχουν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα αλλά και τους ίδιους τους εργαζομένους. Νομίζω ότι και μετά από αυτά τα οποία είπε η κυρία Χάρκινγκ ε, μας βρίσκουν σύμφωνος για την γραμμή του προϋπολογισμού η οποία θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την κοινωνική επιχειρηματικότητα είναι σαφές ότι σήμερα δεν υπάρχει αλλά νομίζω ότι με το χρόνο μπορέσαμε να διαπιστώσουμε ότι ορισμένες ε, ιδέες οι οποίες στην αρχή θεωρήθηκαν ανέφικτες με τον καιρό κατέστησαν εφαρμόσιμες. Να ξεκινήσουμε λοιπόν έστω και με μια πρόκληση για το μέλλον λέγοντας το τι είναι σημαντικό. Υπάρχουν κανόνες, είναι σαφές, είναι αυστηροί κανόνες, είναι επίσης σαφές, αλλά αν δει κανείς το νέο σχέδιο Juncker, το στρατηγικό αυτό σχέδιο, το οποίο θα πρέπει να γίνει δεκτό και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να υπάρξει διαδικασία εκδοσής εγγυήσεων για τις πιστώσεις, Νομίζω ότι μένει πολλά να γίνουν, υπάρχουν οι κανόνες αλλά πολλές φορές υπάρχουν και αποκλήσεις όταν αυτό είναι απαραίτητο. Λοιπόν και εκεί όπου είναι απαραίτητο μπορούμε να φανούμε λίγο πιο τολμήροι. Ευχαριστώ η κυρία Ριμπέιρο έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τη συνάδελφο Βερόνικα Φοντανιέ για μια έκθεση σε ένα θέμα το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την απασχόληση. Πρόκειται για μια ρύθμιση η οποία θα επηρεάσει πάνω από 2 εκατομμύρια επιχειρήσεων που ασχολούνται με τα θέματα αυτά, 14 εκατομμύρια θέσεων εργασίας, 5% περίπου των εργαζομένων. Έτσι θα καταπολεμήσουμε λοιπόν την ανεργία των νέων και την μακρόχρονη ανεργία. Αυτό δίνει την δυνατότητα λοιπόν σε αυτούς που έχουν απομακρυνθεί από την αγορά εργασίας. Οι κοινωνικές αυτές επιχειρήσεις πολλές φορές δεν αναγνωρίζονται νομικά στην Ένωση και αυτό δημιουργεί προβλήματα όταν αναζητούν χρηματοδότηση και τις θέτει σε κίνδυνο. Γι' αυτό λοιπόν και σύμφωνα με τις προτάσεις που έχουν ήδη γίνει, νομίζω ότι θα πρέπει να τονίσουμε τον ρόλο των επιχειρήσεων αυτών και να τις συμπεριλάβουμε ε, στους στόχους σε αιτήσια βάση. Η Επιτροπή έκανε ένα πρώτο βήμα, δημιούργησε μια ειδική μονάδα ε, για τον τομέα αυτό, αλλά χρειάζεται μια μεγαλύτερη ε, θα έλεγα υπογράμμιση και θα πρέπει να δοθεί και μια ξεκάθαρη νομική βάση σε αυτές τις επιχειρήσεις. Μπορούμε λοιπόν να θεωρήσουμε ότι παίζουν ένα σημαντικό ρόλο για να βοηθήσουν την καταπολέμηση της φτώχειας. Thank you. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Φωντανιέ, θέλετε κάτι να προσθέσετε μετά από αυτή τη σύντομη συζήτηση. Να ευχαριστήσω όσους πήραν το λόγο μέχρι τώρα. Να πω ότι θα συμφωνήσω με αυτά τα οποία είπαν και πράγματι θα προσπαθήσουμε να καταλήξουμε στις συμβιβαστικές προτάσεις και θα ξεκινήσουμε ήδη από το απόγευμα. Uh, ευχαριστώ πολύ. Η ψηφοφορία στην απασχόληση θα γίνει στις 15, στην Επιτροπή Απασχόλησης στις 15 Ιουλίου. Σας ευχαριστώ όλους για τη συμμετοχή σας. Η επόμενη συνάντηση την 23η Ιουνίου. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε. Thank you for today.